Good morning, everybody. Um, in spite of the limited appearance of the committee, which is partly due to our EPP staying Helsinki. Καλημέρα. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση λόγω κάποιων συναδέλφων που ήταν ε, στο Ελσίνκι. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση σήμερα. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπορεί να εγκριθεί χωρίς καμία αλλαγή. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση, οπότε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχω κάποιες ανακοινώσεις προς την Επιτροπή. Πρώτον, θα έχουμε ε, μια ημερίδα που θα οργανωθεί για τον εγκέφαλο, για τη νέα προσέγγιση για τις ε, ασθένειες του εγκεφάλου. Θα οργανιστούν από τη Health Working Group με συμπροεδρία Σολεδάδη Καμπεσορουής και Αλός Πέτερλε από 21 Νοεμβρίου ε, στι 21 Νοεμβρίου, συγγνώμη, από τι 10 το πρωί μέχρι τι 12 το μεσημέρι. Και όλα τα μέλη είναι ευπρόσδεκτα. όλα τα μέλη τη ΕΜΒΗ. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες εκτός από εστονικά, λετονικά και ιρλανδικά. Ε, μεταδίδεται σε, με web streaming η συνεδρίαση και τα αρχεία της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Να σας ε, αναφέρω για τις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη μείωση της επίπτωσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Είναι ένα σημαντικό θέμα συζήτησης με τα όργανα. Ο πρώτος άτυπος τρίλογος ε, για την πρόταση για τα πλαστικά μίας χρήσης έλαβε χώρα την 3η 6 Νοεμβρίου στους χώρους του Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων περί των κυρίων στοιχείων των θέσεων των συνομοθετών. Ακολούθησαν εκτενεί συζητήσει για διάφορα ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κατανάλωσης και μείωση στο άρθρο 4, το πράγμα 1, τμήμα α, τους περιορισμούς για την κυκλοφορία στην αγορά, στο άρθρο 5 και το παράρτημα 1 μέρος β αλλά και για την εκτεταμένη ευθύνη παραγωγών, την EPR στο άρθρο 8 και μετά ε, στο παράρτημα 1 τμήμα α και τα ξεχωριστά μέτρα περισυλλογής ε, στο άρθρο 9 και στο παράρτημα 1F. Υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν όλες οι τροπολογίες ε, για να παρασχεθούν κάποιες διευκρινήσεις και να υπάρχει κάποια ευθυγράμμιση σε τεχνικά ζητήματα. Ο δεύτερος τρίλογος για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα έχει προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα στην πρώτη μας ε, συζήτηση σήμερα. Είναι μια κοινή συζήτηση για την υλοποίηση της, ε, για την εφαρμογή της οδηγίας 2928 έκα σχετικά με την ορθολογική χρήση των κυριακών φαρμάκων μαζί με την παρουσίαση της μελέτης της EPRS για την εκτίση εφαρμογής σχετικά με την ορθολογική χρήση των κυριακών φαρμάκων. Η συγητής είναι η Γιούτε Γκίτελαντ, η συγγήτρια, συγγνώμη. Όσον αφορά το πώς θα οργανώσουμε τη συζήτηση τώρα, πρώτα δίνω τον λόγο στην EPRS για να μας κάνουν μια παρουσίαση της μελέτης ε, σε χρόνο 15 λεπτών ε, τόσο χρόνο έχουμε από όσο ξέρω θα χωρίσετε διάφορα ζητήματα εσείς μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά χρόνο που σας δίνουμε για την παρουσίαση της μελέτης EPRS ε, και μετά θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια η οποία βρίσκεται και εδώ μάλιστα, καλώς ορίσατε και στους σκιώδεις στη συνέχεια και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής το επιθυμεί, αλλά και για τα μέλη των ε, Επιτροπών Άγκρη. Πέστε, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και το επιτελείο της για την υποστήριξη που είχαμε ε, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, εξωτερικούς μας ερευνητές, ε, το Arcadia International και το ο τον Ντανιέλ Tron και την Ελέν Γκορνή, στους οποίους και θα δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσουν αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ Μίλα κύριος Ντανιέλ Τράουν. Κυρίες και κύριοι, μαζί με τη συνάδελφο Ελένη Κογνή, ε, θεωρούμε τη βήμα την ευκαιρία που έχουμε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη αυτή ε, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009 128 για την ορθολογική και βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Μετά από τη σύντομη εισαγωγή. Θα σας πούμε τα βασικά ευρήματα και πορίσματα και τέλος θα προχωρήσουμε σε ένα κατάλογο συστάσεων. Η μελέτη έλαβε χώρα από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο φέτος για μια εξπόστ αξιολόγηση ε, της εφαρμογής της οδηγίας. Ε, κοιτάξαμε πώς μεταφέρθηκε, πώς ε, υλοποιήθηκε και πώς επιβλήθηκε ιδιαίτερα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μείωση του κινδύνου και όχι μόνο. Η μεθοδολογία βασίζεται σε μία προσέγγιση δύο επίπεδων. Το πρώτο επίπεδο ήταν να γίνει αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής της ε, οδηγίας χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων ε, ανάλογα με την σκοπιμότητα, αποτελεσματικότητα και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Γενικά ε, κάναμε και μια επισκόπηση της ε, βιβλιογραφίας. Είχαμε δύο πάνελ, ένα για τους ενδιαφερόμενους χρήστες και το άλλο ήταν για τις κρατικές αρχές. Τρία θέματα μας ε, ενδιαφέραν σε τρεις ομάδες ε, να έχουμε δείκτες που μετρούν τον κίνδυνο, να δούμε πώς εφαρμόζεται η οδηγία ε, σε σχέση με τον περιορισμό και την απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Και τέλος μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μελέτη σε σχέση με το πόσιμο νερό και πώς ε, συλλέξαμε τα στοιχεία σε έξι ε, με βάση πάντα τη βιβλιογραφία αλλά και ερωτήσεις που κάναμε στους ενδιαφερόμενους. Πριν σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα θα θέλαμε να κάνουμε δύο εισαγωγικά σχόλια. Πρώτον, να τονίσουμε ότι η οδηγία καλύφθηκε και ένα νέο τομέα πολιτικής που προηγουμένως δεν ρυθμιζόταν. Γι' αυτό τα εθνικά επιχειρησιακά σχέδια ήταν καινούργια για τα περισσότερα κράτη-μέλη. υπάρχει τώρα ένα διάστημα, μια διαφορά φάση ανάμεσα στη στιγμή που εφαρμόστηκε η οδηγία και τα βυθινητά αποτελέσματα. Την τελευταία δεκαετία έχουμε ένα status quo το οποίο έχουμε παρατηρήσει. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και παρελθούσες μελέτες που είχαμε κάνει και είδαμε ότι παρέμειναν σταθερές ε, οι θέσεις και των ενδιαφερομένων των συμφεροντούχων και των κρατικών αρχών την τελευταία δεκαετία. Μετά είδαμε ποιος ήταν ο βαθμός απόκρισης ε, ε, στο ερωτηματολόγιο μας οι ενδιαφερόμενοι φορείς απάντησαν ικανοποιητικά οι κρατικές αρχές μάλλον κάπως απρόθυμα. Ο στόχος τη οδηγία παραμένει ενισχύ και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αλλάξει η νομοθεσία. Πολλοί ΜΚΟ όμως πρότειναν να προσθέσουμε ένα επιπλέον στόχο, δηλαδή να μειώσουμε την εξάρτηση από τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Γιατί θεωρούν οι ΜΚΟ ότι σήμερα δεν εφαρμόζεται αρκετά αποτελεσματικά ο στόχο αυτό. Οι ίδιες ΜΚΟ είπαν ότι ε, πρέπει να συνεχιστούν κάποιες προσπάθειες για την αύξηση της συνοχής, πούμε, η, συνοχή, η νομική συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθεσιών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γενικότερο νομικό πλαίσιο. Στη θεωρία αυτά ισχύουν, αλλά Είναι πολύ αργές οι διαδικασίε έγκριση α πούμε, για τις ουσίε ε, χαμηλού ρίσκου, χαμηλού κινδύνου και την κυκλοφορία του στην αγορά. Το έχουμε δει και σε άλλες εκθέσεις, αυτό ιδιαίτερα. Στην πρόσφατη αξιολόγηση ε, του αντίστοιχου νόμου. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα τώρα, την αποδοτικότητα, έχει γίνει πρόοδος στα περισσότερα κράτη-μέλη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν να εκπαιδεύουν ε, επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα αυτά σχετικά με τους κινδύνους και τον περιορισμό τους. Βέβαια είναι πολύ λίγα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που υπάρχουν σε σχέση με το στόχο μείωση του κινδύνου. Πολύ λίγα είναι τα κράτη-μέλη που έχουν βάλει ποσοτικούς στόχους για τη μείωση της χρήσης ή των ποσοτήτων και τον περιορισμό του κινδύνου. Αυτό έχει να κάνει ιδιαίτερα ε, με την εφαρμογή του άρθρου 15 της οδηγίας για το IPM και δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Και επίσης οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν ε, επαρκώς ε, ακόμα τι σημαίνει το IPM. Αποδοτικότητα εδώ έχουμε πρόβλημα έλλειψης πόρων και οικονομικών και ανθρώπινων για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Με εξαίρεση τη Γαλλία. Επίσης και στη χρηματοδότηση της έρευνας δεν υπάρχουν ε, αρκετοί πόροι, χρηματοδότηση δηλαδή για να εφευρεθούν ε, εναλλακτικοί τρόποι φυτοποστασίας. και συνεχώς μειώνεται το προσωπικό. Τελευταίο κριτήριο στην αξιολόγηση ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εδώ υπάρχει μεγάλη συνένεση μεταξύ των απαντώντων στην έρευνα ότι τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να επιτύχουν κανένα αποτέλεσμα χωρίς την οδηγία. Αν δεν υπήρχε οδηγία δηλαδή αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Επίσης η οδηγία αυξάνει τη συνειδητοποίηση ε, των επαγγελματιών και των κρατών μελών. Αυτά ήταν τα ευρήματα λοιπόν της αξιολόγησης και μετά ε, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, οι δείκτες κινδύνου. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το καιρό ε, προετοιμάζουν το παράρτημα 4 για τους δείκτες της οδηγίας αυτής. Ε, από τη μελέτη οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα ότι υπάρχουν διάφοροι δείκτες που έχουν αναπτυχθεί κατά την περίοδο 2005-2015 και απλή περιγραφική και πιο περίπλοκη ε, ε, για τον υπολογισμό ε, του κινδύνου με βάση κάποια περίπλοκα μοντέλα. Την τελευταία πενταετία όμως έχει χαλαρώσει αυτή η προσπάθεια γιατί περιμένουν να εγκριθούν εναρμονισμένοι δείκτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κακή ποιότητα τα στοιχεία για τη χρήση των φυτοφαρμάκων και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για ε, την ε, κατάρτιση δικτών, ιδιαίτερα εκείνων που αυσίζονται σε μοντέλα. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου σε κάποιους συγκεκριμένου τομεί και οι περιοχές είναι το άρθρο 12 της οδηγίας, αυτός ο περιορισμός ήδη έχει ε, εφαρμοστεί με βάση ε, την, τον αντίστοιχο κανονισμό 1107 του 2009. Ε, και διάφορα κράτη-μέλη έχουν επιβάλει επιπλέον περιορισμού σε κρατικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν απαγορεύσει τη χρήση φυτοφαρμάκων στους δημόσιους χώρους και υπάρχουν και άλλες χώρες που το συζητούν αυτό. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα εθνικά προγράμματα δράσης δεν περιγράφουν ρητά τα μέτρα που παίρνουν ε, να προτιμούν προϊόντα χαμηλού κινδύνου ή βιολογικά μέτρα. Τέλος, τι γίνεται με την παρουσία επικίνδυνων τοξικών χημικών ουσιών στο πόσιμο νερό. Υπάρχουν ευρύτατα συστήματα ελέγχου ε, σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ε, για όλες τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Επίσης, ε, με βάση το τοξικολογικό προφίλ κάθε ουσίας ε, υπάρχουν και κάποιες περιοχές απομόνωσης. Τι γίνεται με τις μελέτες τώρα, τις κοινωνικονομικές και τις περιβαλλοντικές ε, για την ποιότητα του ποσίμου ύδατος. Πραγματικά χρειάζονται ε, τέτοιες μελέτες ευρύτερες γιατί σήμερα δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία. Σήμερα μετράνε μόνο τις ουσίες και τις ωριακές τιμές και αν αυτές ε, είναι στα φυσιολογικά επίπεδα ή όχι. Συστάσεις λοιπόν. Προτείνουμε τρία αιώνιδων συστάσεις. Πρώτον, γενικής φύσεως για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και η σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Εδώ συστήνουμε στις κρατικές αρχές να πρωταγωνιστήσουν ε, στις εξελίξεις. Δηλαδή να μην περιορίζονται μόνο στο να ελέγχουν κάποιες δραστηριότητε, αλλά να είναι και η κινητήρια δύναμη ε, για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Τα κράτη-μέλη επίση θα πρέπει να επιζητούν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών, ας πούμε Υπουργεία Περιβάλλοντος, Υπουργεία Γεωργίας κτλ. Και, τα οι κρατικές αρχές να λειτουργούν συντονιστικά. In addition... Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών και να ενθαρρυνθεί. With respect to the revision... Σε σχέση με την αναθεώρηση των ΝΑΠ, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν ε, ποσοτικούς στόχους που σήμερα δεν υπάρχουν αυτά και επίσης να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και χρονική δράση με δράση και σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμα από την οδηγία, αλλά που μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της υλοποίηση. Άλλες συστάσεις πέρα από τις γενικές ε, για καλύτερη εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυτοφαρμάκων, IPM. Θα πρέπει πρώτα να το καταλάβουν αυτό οι εθνικές αρχές, ότι χρειάζεται χρόνο, αλλά και το κοινό για, να αλλάξει στον τύπο καλλιεργειών σε μια χώρα, αυτό είναι μια υπόθεση μακράς πνοής ε, και σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι το απλό και το βραχυπρόθεσμο. Και χρειάζεται προσέγγιση για μια ε, ε διαρθρωμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση ε, για τα φυτοφάρμακα ανάλογα με το προϊόν. Κάτι που είναι καλό ας πούμε, για τις δομάτες στην Ισπανία δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάπου αλλού. Είναι αυτά τα μέτρα ειδικά ανακαλλιέργεια και ένα χώρο Για παράδειγμα, οι ομάδες επιχειρησιακές που έχουν δημιουργηθεί είναι μια καλή αφετηρία για να υπάρχουν διάφορες και πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών κλπ. όπως το Eranet ε, είναι μια καλή ε, επίσης πρωτοβουλία. Και τέλος, ε, πάντα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτοφαρμάκων, δεν έχουν γίνει ακόμα αρκετές προσπάθειες για την έρευνα και την ανάπτυξη και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το προωθούν και χρειάζονται και ανεξάρτητες υπηρεσίες παροχής συμβουλών για να ενημερώνονται σωστά οι παραγωγοί ή οι γεωργοί Και επειδή είναι υψηλό το κόστο αυτό θα πρέπει να αντισταθμίζεται με επιδοτήσεις, με ασφάλειες ε, και με κίνητρα από τις αγορές και τις χρηματαγορές για να γίνει αυτή η μετάβαση προς τη ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτοφαρμάκων. Επίσης να αναπτυχθούν περισσότερο οι δείκτε που βασίζονται σε μοντέλα. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, καταβάλουν περισσότερε προσπάθειες προ την κατεύθυνση αυτή και να μην έχουν απλώς έτσι περιγραφικούς δείκτες και γενικής φέσης. Και ένα τελευταίο, χωρίς να είναι το λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να κάνουν φιλόδοξες προσπάθειες στα κράτη-μέλη για να συλλέγουν στοιχεία αξιόπιστα για ε, τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Εδώ τελειώνει η σύντομη παρουσίαση μας για τη μελέτη. Σας ε, καλούμε να τη διαβάσετε σε λεπτομέρειες, ε, γιατί περιλαμβάνουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση θα είχατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που ε, τηρήσατε και το χρόνο ομιλία. Και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κουτελάντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και για την εξαιρετική έκθεση και την παρουσίαση που ακούσαμε σήμερα από το EPRM. Θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μου και θα επανέλθω και σε πολλά από αυτά που ανέφερε το EPRS σχετικά με την ε, έκθεσή μου. Ε, η αηφόρος ε, χρήση, μάλλον η οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από το 2012 και σκοπό έχει να διασφαλίσει την αηφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Έτσι έχουμε την ε, ολοκληρωμένη διαχείριση φυτοφαρμάκων και είναι ε, απαραίτητο αυτό ώστε η Ευρώπη να στραφεί προς μια πιο αηφόρο γεωργία που να μπορεί να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο παραγωγής τροφίμων ε, αλλά ταυτόχρονα με αφαίρεση των ε, επιβλαγών ουσιών από το έδαφος. Όσον, αφορώ, όσον αφορά την αδειοδότηση των ε, φυτοφαρμακών στην Ευρώπη, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε πώς εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη την οδηγία αυτή. Και έχω βασίσει την έκθεσή μου και τις εργασίες μου ε, πάνω στο σχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, καθώς και στην επιστημονική μελέτη του ε, EPRS που μόλις ακούσαμε. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για τη μελέτη αυτή. Έχουμε σαφή εικόνα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Ε, παρότι κάποια κράτη-μέλη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, ε, το γενικό επίπεδο εφαρμογής ε, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση και μάλιστα αντί για να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη, έχουμε δει αύξηση από τα μέσα της δεκαετία του 90 και ενώ υπάρχουν νέα φυτοφάρμακα στην αγορά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χαμηλή δόση, η χρήση κατά μέσο όρο δεν μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Φυσικά η χρήση των φυτοφαρμάκων παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωργική παραγωγή της Ευρώπης, διατηρώντας την υγεία των φυτών. Ωστόσο, είναι γεγονό ότι μπορούν να έχουν αρνητικέ επιπτώσει τα φυτοφάρμακα στην ανθρώπινη υγεία, επηρεάζουν δε και το οικοσύστημα και ε, συμβάλλουν στη μείωση της βιοπικιλότητας και βλέπουμε ιδιαίτερα μεγάλη μείωση ε, του πληθυσμού των εντόμων. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για πολλούς λόγους. Φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον να προστατεύονται από επικίνδυνα χημικά. Τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ενώ τα κατάλοιπα στις ζωοτροφές ε, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και μπορούν επίσης να εισέλθουν στην ε, αλυσίδα τροφίμων. Βρίσκω απαράδεκτο το ότι ακόμη υπάρχουν φυτοφάρμακα που ε, υποπτευόμαστε ότι μπορούν να προκαλέσουν ενδοκρινικέ διαταραχέ, ε, και παρόλα αυτά διατίθενται ε, στην Ευρώπη. Αυτές ε, τις ουσίες θα πρέπει να τις εντοπίσουμε σύμφωνα με τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν πρόσφατα και δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά τέτοια φυτοφάρμακα. Η μη αηφόρος χρήση των ε, φυτοφαρμάκων ε, είναι επιβλαβής και για την παραγωγή των τροφίμων, διότι γνωρίζουμε ότι η παραγωγή των τροφίμων εξαρτάται από την επικονίαση από τα έντομα. Όταν λοιπόν αυτά τα έντομα ε, πεθαίνουν λόγω της μη βιώσιμη χρήσης των χημικών, αυτό είναι πολύ ανισχυτικό και για την Ευρώπη και για όλον τον κόσμο. Μάλιστα, είναι όλο και πιο σαφές ότι αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση θα πρέπει να αποτρέψουμε την κατάρρευση των οικοσυστημάτων και την απώλεια βιοπικιλότητας. Μια πρόσφατη ε, μελέτη του WWF έδειξε ότι το 60% των ε, ε, θηλαστικών ερπετών ε, και ε, εντόμων ε, έχει εξαφανιστεί από, το, από τη δεκαετία του 1970. Βλέπουμε επίση ότι ο πληθυσμό των εντόμων έχει μειωθεί κατά 75% στη Γερμανία τα τελευταία 30 χρόνια και στι δύο περιπτώσει οι επιστήμονε αναφέρουν την χρήση των φυτοφαρμάκων ω μία από τι αιτίε για αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα. Για να είναι πιο βιώσιμη η γεωργία όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, χρήση φυτοφαρμάκων στα σημερινά επίπεδα. Ε, είναι το βασικό μέσο για τον έλεγχο των ε, επιπλοκών οργανισμών, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. διότι βλέπουμε και αύξηση της ανθεκτικότητας ε, των επιβλαβών οργανισμών και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ε, της οδηγίας, κάτι που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Ε, έχουμε, κάποια, ε, έχουμε παρατηρήσει κάποια πρόοδο όσον αφορά τον εξοπλισμό ψεκασμού. Έχουν δοθεί οδηγίες για, την, ε, για τις καλύτερες μεθόδους ψεκασμού, ωστόσο ε, πολύ περιορισμένη η χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών ε, έχει υπάρξει κάτι που είναι απαραίτητο. Επίσης, δεν υπάρχουν σαφείς και ποσοτικοί στόχοι στα εθνικά σχέδια δράσης. 21 ε, κράτη-μέλη έχουν ε, θέσει στόχους. Ε, όσον αφορά τον κίνδυνο αλλά και τη μείωση της χρήσης, μόνο τέσσερα κράτη-μέλη τελικά έχουν στόχους μείωσης του κινδύνου, κάτι που σίγουρα δεν αρκεί. Αυτή η έλλειψη ποσοτικών στόχων μετρήσεων και χρονοδιαγραμμάτων για τις διάφορες περιοχές σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, τα περισσότερα σχέδια δράσης δεν αναφέρουν πώς θα επιτευθούν αυτοί οι στόχοι και πώς θα μετρηθούν. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει ούτε πρόοδος ε, στην, όσον αφορά την ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών που αποτελεί θεμελιώδη λίθο αυτής της οδηγίας και που στόχο έχει να περιορίσει την χρήση φυτοφαρμάκων σε επίπεδα επιτρεπτά όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν ε, να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μεθόδους για να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες. Δυστυχώς ε, τα κράτη-μέλη σήμερα δεν έχουν εφαρμόσει πλήρω ε, τι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, αλλά θεωρούν ότι αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι μάλλον μέσω κατάρτιση των γεωργών, ούτε έχουν τρόπο αξιολόγηση τη συμμόρφωση με τι αρχέ αυτέ. Υπάρχουν ε, τεράστιες δυνατότητες στην ολοκληρωμένη διαχείριση όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή την εργαλειοθήκη όσο γίνεται πιο σύντομα. Ένας τρόπος να αυξηθεί η χρήση των πρακτικών της ολοκληρωμένης διαχείρισης ε, του IPM είναι να υπάρχει ε, πολλαπλή συμμόρφωση ε, όσον αφορά αυτήν την οδηγία και την οδηγία άμεσων ενισχύσεων. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικά κίνητρα για τη χρήση της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στην έκθεσή μου διαπιστώνεται ότι υπάρχει ε, επιτακτική ανάγκη να ε, αυξηθεί η προσβασιμότητα σε εναλλακτικέ ε, λύσεις όπως είναι τα προϊόντα φυτοπροστασία χαμηλού κινδύνου. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε βιώσιμη γεωργία και για να διευρύνουμε την εργαλειοθήκη των γεωργών, αυξάνοντας τις δυνατότητες που έχουν για φυτοπροστασία. Γνωρίζουμε ότι πολλοί γεωργοί χρησιμοποιούν χημικά, παραδοσιακά χημικά μέσα φυτοπροστασίας αντί να δοκιμάζουν νέες μεθόδους. Δεν φταίνε οι γεωργοί σε αυτό, διότι πιο πολύ τους ενδιαφέρει η καλλιέργεια. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να μειώνουν οι γεωργοί την χρήση φυτοφαρμάκων και να μεταβούν σε μη χημικές λύσεις. Και Γι' αυτό είναι απαραίτητη η έρευνα και ανάπτυξη για να αναπτυχθούν εναλλακτικέ λύσεις προστασίας ε, κατά επιβλαβών οργανισμών, ε, ε, παρόντων και μελλοντικών, κάτι που θα μειώσει τη χρήση των μέσων φυτοπροστασίας και να έχουμε νέους τρόπους δράσης. Άλλο βασικό συμπέρασμα έχει να κάνει με τους εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου παρά την ε, σαφή υποχρέωση ε, στο άρθρο 15 της οδηγίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη δεν έχει εκπονήσει τέτοιους δείκτες που θα δείχνουν ότι που θα επιτρέπουν την σωστή μέτρηση των ε, αποτελεσμάτων και γι' αυτό ε, απομένουν να γίνουν περισσότερα στον τομέα αυτών. Και τέλος, καθότι ε, τέτοιες εκθέσεις ε, εφαρμογής ε, είναι κάπως περιορισμένες όσον αφορά το εύρος τους, θα υποβάλω επιπλέον τροπολογίες. Προσβλέπω στις τροπολογίες των συναδέρφων την επόμενη εβδομάδα και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές για να πετύχουμε ισορροπημένο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή ορισμένοι συναδελφοί δεν βρίσκονται εδώ, πάμε στην επόμενη, στον επόμενο σκιοδησίγητη, τον κύριο Γιάννη Χέταμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΙΟΤΕ για την έκθεση της ε, και προσβλέπω σε μια εξαιρετική συνεργασία και σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν θα επαναλάβω όσα είπε η συγγήτρια αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα ήθελα να εστιαστώ ε, ε, όπως θα κάνουμε στις τροπολογίες μας ως Άλντε. Θέλουμε να έχουμε κάποιες εναλλακτικέ ε, χαμηλή κινδύνου, το λέμε εδώ διαρκώς ε, στο Κοινοβούλιο να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες εξουσιοδότησης ταχύτερες ενδεχομένως για, τις, για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών επίσης. Αυτό είναι σημαντικό πρέπει να ενταχθεί στη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ισοδύναμο του greening. Και αυτό ήθελα να τονίσω. Πολλές φορές στην κοινή γεωργική πολιτική έχουμε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τα μέτρα greening. Είναι μια γενική προσέγγιση ε, για όλα. Εγώ θα ήθελα ε, μια πιο συντονισμένη, ε, ε, στοχευμένη προσέγγιση βάσει στόχων. Ήθελα λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη αναλογικότητα των οικολογικών συστημάτων στη γεωργική πολιτική όπου εντάσσεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτά τα eco-schemes, τα οικολογικά προγράμματα να είναι ευρύτερα και βάσει αυτής της ε, προσέγγισης που έχουμε χαμηλού κινδύνου. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει και η ολοκληρωμένη ε, διαχείριση επιβλαβών οργανισμών σε σχέση με τις διάφορες καινοτομίες τεχνολογικές ε, και οικολογικές. Είναι ένας πολύ καλός συνδυασμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών και ενδεχομένως την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών Ορισμένε φορέ ω τελευταία λύση, ω εσχατή λύση, χρειάζεται κανεί χημικά ή οργανικές ε, ουσίες για την προστασία ε, των χωραφιών. Και μετά πρέπει να δούμε αν χρησιμοποιήσουμε πολύ λίγη δραστική ουσία, ε, πολύ μικρή ποσότητα κάποιας δραστικής ουσίας, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος σε σχέση με το αν χρησιμοποιούμε υψηλής επικινδυνότητας ουσίες. Ε, δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε πολλέ ουσίε χαμηλού κινδύνου, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ότι αν χρησιμοποιούμε λίγε ουσίε υψηλού κινδύνου. Οπότε πρέπει να δούμε πρακτικά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ε, αν χρησιμοποιούνται πολύ μικρέ δόσει ε, πολύ αποτελεσματικών ουσιών υψηλού κινδύνου, μπορεί αυτό να είναι καλύτερο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η βιωσιμότητα και τα φυτοφάρμακα ε, δεν χωράνε στην ίδια πρόταση. Ε, κανονικά δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε στην ίδια πρόταση. Ε, τα φυτοφάρμακα είναι χαρακτηριστικό για την εντατική μέθοδο με την οποία παράγουμε τα τρόφιμά μας θα πρέπει δηλαδή να αυξάνεται η παραγωγή όσο περισσότερο γίνεται με το μεγαλύτερο δυνατό, μικρότερο δυνατό κόστος, εξού και τα φυτοφάρμακα. Αυτό έχει επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, για το περιβάλλον, το πόσιμο νερό, την υγεία των ζώων και τη βιοποικιλότητα. Αυτό αφορά όμως και την παραγωγή τροφίμων. Ε, γιατί τα έντομα της επικονίασης ε, ε, σιγά σιγά αφανίζονται και πού είναι εδώ η βιωσιμότητα και παρά τον, την επικεφαλίδα η συγγήτρια έκανε μια καλή έκθεση και μιλά για την αρχή της προφύλαξης και τη θεωρία φετηρία. Είναι σημαντικό. Επικρίνει επίσης τα κράτη-μέλη ε, στην εφαρμογή, ζητάει στόχους πραγματικούς και μετρήσιμους και απαγόρευση ουσιών ε, που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές ε, ή είναι επικίνδυνα χημικά για τον άνθρωπο. Θα πρέπει να περάσουμε όμως προς μια βιώσιμη παραγωγή και να μας ενδιαφέρει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και με τους άλλους και οδησηγητές για να βγάλουμε μια βιώσιμη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο... και στα επιπλέον ε, μέλη της Επιτροπής Τσάγκρη, της ΠΕΣΤΑ, αν υπάρχουν εδώ. Η κυρία είναι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ε, Γιούτε Γκιουτελάντα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η παρουσίαση που μας έκανε. Μας έδειξε ότι επήγει η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Να σας αναφέρω μια μελέτη που κάναμε εμείς ως πράσινη με πάνω από 150 εθελοντές σε 6 χώρες της Ευρώπης και δοκιμάσαμε 30 φυτοφάρμακα. Ω δείγμα πήραμε τα μαλλιά. Και ξέρετε, τα μαλλιά έχουν κάποιο ενδιαφέρον, διότι ένα ε, εκατοστό παρουσιάζει την επίδραση σε διάστημα ενό μήνα. Και βρήκαμε ότι σε δύο στου τρει Ευρωπαίου έχουμε μολυνθεί. Έχουμε φυτοφάρμακα πρακτικά κατά μέσο όρο πάνω από 60% ε, στο πάνω, σε πάνω από 60% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που δοκιμάσαμε. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ σοβαρή. Δεν μπορούμε να πούμε αν ε, ένα σωρό κόσμο δεν έχει μολυνθεί, ακόμη και αν τρώει κανεί βιολογικά και πάλι μολύνεται. Και αυτό που μα κάνει έκπληξη είναι να δούμε τον τύπο των μολύνσεων που έχουμε. Έχουμε φιμπρονίλ για παράδειγμα, το οποίο έχει απαγορευτεί στη Γεωργία από το 2017. Στη δική σα όμω έκθεση ε, του IPRS ε, θα ήθελα να μας λέτε ότι βλέπετε τη μόλυνση αυτή όχι μόνο τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στη, στη Γεωργία αλλά και τα βιοκτώνα διότι η δραστική ουσία φιπρονίλ χρησιμοποιείται στα βιοκτώνα. Κάναμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ ενός πατέρα που είχε μια μόλυνση 1 το παιδί είχε τριπλάσια διότι και οι γάτες ε, που υπήρχαν στο σπίτι όλα αυτά επηρεάζουν ε, την υγεία. Και μετά έχουμε το το περιφός το οποίο έχει απαγορευτεί αλλά που το βρίσκουμε για παράδειγμα στη Γαλλία στα, στις τρίχες ε, και αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Αυτό που θέλω να δω λοιπόν στην έκθεσή σας και μετά θα κλείσω. Ε, ξαναδιαβάστε την έκθεσή σας. Ε, ξαναδιαβάστε την έκθεση. Έχει γίνει, την έκθεσή μας έγινε από ένα εργαστήριο στο Στρασβούργο και παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μόλυνσης. Μιλάμε για εφήβους 10 έως 17 ετών ε, ομάδα ηλικιακή που παρουσιάζει την υψηλότερη μόλυνση. Μιλάτε για τις ε, επιπτώσεις στην υγεία και τελικά να έρχεται κανεί ποια είναι η εικόνα της Ευρώπης Ενό χώρου που δεν προστατεύει τους πολίτες της και την υγεία τους. Έχουμε εκατοντάδε φυτοφάρμακα, φυτοφάρμακα που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και κυκλοφορούν στην αγορά. Φυτοφάρμακα όπω το, ε, το περιφώς που κυκλοφορούν στην αγορά που τα βρίσκουμε σε δείγματα, διάφορα καρκινογόνα που τα βρίσκουμε σε διάφορα δείγματα, θέλετε να σκοτώσετε του Ευρωπαίους πολίτες. Και σας βρίσκω υπερβολικά χαλαρού στα όσα προτείνετε. Θα έπρεπε να είχατε πάει και να είχατε πει πρέπει να απαγορέψουμε τα καρκινογόνα, τα μεταλλαξιογόνα, τους ενδροκρινικούς διαταράκτες με κατεπήγουσα διαδικασία. Το δεύτερον θα ήθελα να ε, στραφείτε κατά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έπρεπε να θεσπίσει τα κριτήρια. Είδατε πόσο έχει καθυστερήσει μέχρι να θεσπίσει αυτά τα κριτήρια. Και τώρα έχουμε τα κριτήρια και μετά λένε Α, θα ελαχιστοποιήσουμε του κινδύνου που σχετίζονται με του ενδοκρινικού διαταράκτε. Μα πρέπει να του απαγορέψετε του ενδοκρινικού διαταράκτε. Η δύναμη τη Ευρώπη, αν υπάρχει, και ξέρετε, εμεί η οικολογία είμαστε υπέρ τη Ευρώπη. Η Ευρώπη, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει να γυρνάει και να λέει Εμεί προστατεύουμε την υγεία των πολιτών μα καλύτερα από όλου σα. Εγώ είμαι. Ε, έχετε την... πρέπει να υπάρχει μια διακυβέρνηση. Λέτε, α ναι, κάποιες χώρες ε, κάνουν κάποια μείωση όπως η Γαλλία. Και εγώ Γαλλίδα είμαι. Εδώ και χρόνια λέμε στους Γιώργους πρέπει να μειώσετε την κατανάλωση φυτοφαρμάκων και τι παρατηρούμε το 2017, αύξηση της χρήση των φυτοφαρμάκων. Είχαμε μιλήσει ε, με το σχέδιο Εκοφυτό για μείωση κατά 50% της χρήσης των φυτοφαρμάκων μέχρι το 2025 και δεν είναι, έχουμε, βλέπουμε διαρκή αύξηση. Γιατί δεν φταίνε οι αγρότες. Τα συνδικάτα επιβάλλουν στους γεωργού να χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα γιατί διότι σχετίζονται άμεσα με τα κέντρα ε, πώληση των ε, φυτοφαρμάκων. Ε, και να μιλήσετε για την κοινή γεωργική πολιτική. Πώς θα δεχτούμε μια κοινή γεωργική πολιτική που ευνοεί την εντατική γεωργία. Εντατική γεωργία σημαίνει χρήση φυτοφαρμάκων για αυτού τους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ότι η εκθέσή σας, ναι, κάνει αυτή τη διαπίστωση, δεν ε, είναι όμως καθόλου επιθετική. Θα μα κάνει να πεθάνουμε όλοι σιγά σιγά είναι επίγον το ζήτημα αυτό της υγείας. Έχουμε παραμορφώσει ε, επιδημία καρκίνων και εσείς κάθεστε χαλαροί και λέτε ναι κάποια κράτη θα έπρεπε να κάνουν κάποιες μειώσεις. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Πρέπει να πείτε πρέπει να απαγορεύσουμε ε, ε, τάδε και τάδε φυτοφάρμακο μέχρι το 2020 να γίνει έρευνα, να έχουμε καινοτομία για πιο, λιγότερο τοξικά προϊόντα. Ξέρετε κάτι, η Ευρώπη πραγματικά με κάνει να ντρέπομαι όταν βλέπω ότι εξακολουθεί να αυξάνεται η χρήση των φυτοφαρμάκων στη γεωργία μας και μιλάμε μετά για βιώσιμη γεωργία. Βιώσιμη για ποιον, για την βιομηχανία χημικών, ναι. Αυτό ναι, πράγματι υπερασπίζεστε και στηρίζετε την βιομηχανία χημικών. Τώρα, είναι πολύ καλή η έκθεση τη συναδέλφου θεωρώ, αλλά δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε περισσότερα. Έχουμε επίγον υγειονομικό θέμα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Και δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να ζητούν το λόγο. Ο κύριος Χάιτεμα, ε, μια ε, σύντομη ερώτηση. Ε, προς την προηγούμενη ομιλήτρια, θα απαγορεύατε και το ενόπνευμα, δηλαδή. Σύντομη απάντηση για τη σύντομη ερώτηση η απαγόρευση του ενοπνεύματος, τι σημαίνει. Αν πίνεις ένα ποτηράκι την ημέρα, έχει ανταξιδωτικά που είναι καλό για την υγεία. Φυσικά θα πρέπει να απαγορευτεί το ενόπνευμα για τις εγγύους. Αλλά δεν ε, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι πίνοντας ένα ποτήρι ενόπνευμα τη μέρα θα πεθάνετε. Ενώ αν πάρεις κλορ, ή προπιναζόλη και τα λοιπά, θα δείτε σε λίγα χρόνια πώς θα είσαστε να κλείσει αυτή η συζήτηση. Και αν υπάρχει πρόβλημα με το ενόπνευμα, δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ σχετικό με το θέμα μας αυτό που λέτε. Ο κύριος Μπάλτσο, τελευταίος, όμως, για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη απάντηση σε αυτή την κακή ερώτηση, κατά τα άλλα. Στην περίπτωση του ενόπνευματος, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επιλέγει και να αποφασίζει αν θα πιει ή αν δεν θα πιει. Στα φυτοφάρμακα δεν σε ρωτάνε. Είναι ε, επικίνδυνες ουσίες για την υγεία. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιλέξει. Είναι τεράστια διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος ενδιαφέρεται να τον καλέσω για καμιά μπερίτσα να συζητήσουμε πίνοντας ένα ποτηράκι. Α, συνεχίζει τη συζήτηση. Η κυρία Κάντενμπαχ. Έτσι, έχει φουντώσει η συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Η κυρία Κάντενμπαχ από μια χώρα που είναι γνωστή και φημισμένη για το καλό της κρασί. Εγώ δεν θέλω γενικά να απαγορευτεί το ενόπνευμα. Πάρα πολύ σύντομα, σε σχέση με αυτό που ακούσαμε προηγουμένως για την κατάσταση στην Αυστρία λίγο να σας πω μερικά πράγματα, μια που έχουμε και την Προεδρία του Συμβουλίου και σε πολλούς τομείς ελπίζουμε να είμαστε και υπόδειγμα, όχι σε όλα βέβαια. Ε, παρόλο που ο αριθμός των βιολογικών καλλιεργειών αυξάνεται και σε επιφάνεια στην Αυστρία ε, και μειώνεται ε, η κλασική ε, γεωργία, δεν μειώνεται ο συνολικός αριθμός και τα ποσά των φαρμάκων. Και από τις εκθέσεις βλέπουμε ότι από την αρχή της δεκαετίας του 90 παραμένει σταθερή η ποσότητα που καταναλώνεται. Άρα ε, ε, αυτό τι σημαίνει, ότι στην ε, συμβατική γεωργία έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων, παρόλο που από τη δεκαετία του 90 έχουμε ένα ευρύ πρόγραμμα αντικατάσταση των καλλιεργίων. Παρόλη την κατάρτιση, παρόλη την αλλαγή, δεν έχουμε καθόλου βιώσιμη εξέλιξη, αλλά επικίνδυνη εντατικοποίηση στην Αυστριακή Γεωργία και Φοβάμαι ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την Αυστρία, αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κύριο Σάουν Γκρίφιθ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και το EPRS για την παρουσίαση της μελέτης του. Νομίζω ότι η περίληψη, η σύνοψη των παρουσιάσεων είναι ότι η νομοθεσία είναι κατάλληλη. Ε, υπάρχουν όμως κάποια θέματα όσον αφορά την εφαρμογή. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε κράτη-μέλη, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τις ε, δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω σχετικά με κάποιες από τις δράσεις που έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αυτή τη στιγμή. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια δράσης. Έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα κράτη-μέλη λέγοντας ότι χρειαζόμαστε και περιμένουμε βελτίωση των εθνικών σχεδίων δράσης. Περιμένουμε πιο φιλόδοξους στόχους πιο πολλούς ποσοτικοποιημένους εδίκτες ε, για να μπορέσουμε να ε, ε, καταδείξουμε την επίτευξη των στόχων αυτών. Αναθεωρούν λοιπόν τα κράτη-μέλη τα εθνικά σχέδια δράσης Περιμένουμε τα τελευταία σχέδια δράσης μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα τα επαναξιολογήσουμε και θα εκπονήσουμε περαιτέρω έκθεση που θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο του χρόνου που θα δείχνουν κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει τις συστάσεις μας. Το θέμα του εναρμονισμένου δίκτυ κινδύνου αναφέρθηκε και στις δύο παρουσιάσεις. Αυτή τη στιγμή Έχουμε εκπονήσει έναν τέτοιο δίκτυ, συζητιέται με τα κράτη-μέλη στην ε, ομάδα εργασίας ε, για την ε, βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, όπως συζητιέται σήμερα. Έχει περάσει από διεπηρεσιακή διαβούλευση. Η πολιτική διαβούλευση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και περιμένουμε ψηφοφορία στην Μόνιμη Επιτροπή τον Ιανουάριο. Και κατόπιν θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν τώρα πια έναν τέτοιο δείκτη. Και προσπαθούμε να πετύχουμε τη συμφωνία των κρατών μελών πάνω στον δείκτη αυτών. Αναφέρθηκε η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών ε, και τα ε, μετρήσιμα κριτήρια. Στην ε, αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής έχει αναφερθεί η εισαγωγή της ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών. Για κάτι τέτοιο όπως χρειαζόμαστε μετρήσιμα κριτήρια, ώστε ε, οι γεωργοί να μπορούν να αξιολογηθούν όσον αφορά το θέμα αυτό. Το 2019 λοιπόν στόχο μας είναι να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουμε τέτοια κριτήρια και να δείξουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Έχουμε και το CIPM όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση. Έχουμε προβλέψει μια σειρά προγράμματων κατάρτισης στα κράτη-μέλη που θα ξεκινήσουν ε, φέτος τον Δεκέμβρη, όπου θα γίνουν ε, επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις για να δείξουμε στους γεωργούς πώς να τη χρησιμοποιούν και έχουμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα ε, συνεδριάσει αρχές του επόμενου χρόνου για να καταλήξει σε συμπέρασμα όσον αφορά τα κριτήρια. Κάθε κράτο μέλο πρέπει να έχει μια υπηρεσία παροχή συμβουλών στι εκμεταλλεύσεις, η οποία θα δίνει και συμβουλές όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση. Πρέπει λοιπόν πέρα από τα κριτήρια να φροντίσουμε να υπάρχει και ένας μηχανισμός όπου να μεταφέρει ε, τις ε, μεθόδους αυτές ε, στους ε, γεωργούς. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου και της περιπλοκότητας του θέματος θα κλείσω εδώ. Πάντως συμμεριζόμαστε ε, την ε, την προσήλωση όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων χαμηλού κινδύνου. Έχουμε μια ομάδα εργασία για τον βιοέλεγχο, που θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την διαθεσιμότητα και χρήση των προϊόντων χαμηλού κινδύνου. Επίσης, θα ήθελα να εξηγήσω ότι ο δείκτης που εκπονούμε αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Βασίζεται λοιπόν στις πωλήσει ε, φυτοφαρμάκων, ε, αλλά με ένα ποσοστό διόρθωσης με βάση τον κίνδυνο του φυτοφαρμάκου. Ε, εάν χρησιμοποιεί κανείς λοιπόν φυτοφάρμακο υψηλού κινδύνου, τότε έχει μεγαλύτερο βάρος από ότι ένα φυτοφάρμακο χαμηλού κινδύνου. Ε, ε, ε, αξιολογεί λοιπόν όχι μόνο, εξετάζει όχι μόνο τις ποσότητες αλλά και τον κίνδυνο των φυτοφαρμάκων ο δείχτης αυτός. Σας... Ευχαριστούμε πολύ. Σας δίνω τώρα το λόγο, δίνω το λόγο στην υπηρέσα για μια αντίδραση σε σχέση με τη συζήτηση και την πρόταση της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Με όλες αυτές τις παρατηρήσεις ε, δεν έχω... Άκουσα πολλές παρατηρήσεις, αλλά δεν σημειώσω πολλές ερωτήσεις. Ε, με ερώτηση της κυρίας Ρεβαζή ε, έκανε διάφορα σχόλια όσον αφορά τις ανεπαρκείς φιλοδοξίες στα συμπεράσματα της εκθεσή μας για το ζήτημα της μόλυνσης, της απαγόρευσης των επικίνδυνων προϊόντων και, των δικτών, και τους δείκτες κινδύνου που ανέφερε. Εμείς πραγματοποιήσαμε μια μελέτη ως παρατηρητές αφορά μια οδηγία, ένα νομικό πλαίσιο ε, σε σχέση με τη χρήση των φυτοφαρμάκων ή η απαγορευση των επικίνδυνων προϊόντων ε, Θεσπίστε από τον κανονισμό 1107 για την έγκριση των ε, φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οπότε δεν ενέπιπτε η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της δικής μας μελέτης. Εμείς απλά εξετάσαμε τη χρήση και ως παρατηρητές ε, εποπτεύσαμε την ε, υλοποίηση, την εφαρμογή της οδηγίας και ε, την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία. Και συμπεράναμε μεταξύ άλλων ότι ένα από τα σημεία κλειδιά αυτής της οδηγίας είναι ότι το θέμα δεν είναι η καινοτομία ή έρευνα, είναι ότι δεν έχουμε αρκετά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόθεση των εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης των εναλλακτικών. Αλλά αυτές οι εναλλακτικέ πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει εργαλεία τα οποία θα αντικαταστήσουν τα ε, χημικά προϊόντα, αλλά δεν υπάρχουν απαραίτητα αυτά τα υποκατάστατα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν αυτά τα εργαλεία. Πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτό χρειάζεται χρόνο. Αυτό είναι το βασικό σχόλιο που ήθελα να κάνω σε σχέση με τα όσα ακούσαμε από την κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και την EPRS για τις παρουσιάσεις τους καθώς επίσης και για τη μελέτη. Ήταν πολύτιμη, πολύ χρήσιμη για μένα. Μου δίνει κουράγιο η συζήτηση που γίνεται εδώ στην Επιτροπή σήμερα. Ε, αισθάνομαι την υποστήριξη από πολλούς συναδέλφους ε, για να δείξω φιλοδοξία για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Να τα λάβουμε όλα αυτά πολύ στα σοβαρά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενδυναμώσουμε την έκθεση αυτή, ώστε αυτή να βοηθήσει στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής προσθέτοντας και εργαλεία αναγκαία για ένα πιο υγιεινό και πιο φιλικό περιβαλλοντικά μέλλον. Εγώ ανησυχώ. Παρατηρούμε ε, θάνατο πολλών εντόμων από την εντατική χρήση φυτοφαρμάκων και εγώ ίδια ανησυχώ ιδιαίτερα όταν ακούω ε, να εξαφανίζονται και άλλα ε, ζώα, να πλήττεται ολόκληρο το οικοσύστημα από τη μη βιώσιμη χρήση που παρατηρείται σήμερα. Ανησυχώ λοιπόν και μου δίνει κουράγιο η συζήτηση εδώ σήμερα ε, με τους συναδέλφους οι οποίοι εκφράζουν και ανησυχίες για την ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ε, όταν λένε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την εξαιρετική συζήτηση σήμερα. Αποκόμισα πολλά και αναμένω τις τροπολογίες σας και τη συζήτηση με τους κοιοδησίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του θέματος, τροπολογία της ε, ε, προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 30 Νοεμβρίου 11 21-23 Ιανουαρίου ψηφοφορία στην ΕΜΒΗ. Συγγνώμη, 14 Νοεμβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το Φεβρουαρίου του 2019. Ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και πάμε στο επόμενο σημείο. Έκθεση εφαρμογή σχετικά με τον κανονισμό 1 του 2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κάριν Κάντεμπαχ. Σας δίνω λοιπόν κατευθείαν το λόγο. Κυρία Κάντεμπαχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τώρα εδώ μήπως θα ήταν καλύτερο να ε, ακούσουμε σύντομα την ε, τοποθέτηση της υπηρεσίας ε, μελετών, το EPRS, να μας παρουσιάσει τη μελέτη ή να αρχίσω εγώ με την έκθεση αμέσως, πώς θέλετε. Okay. Then... I think that we should start. I, I, I'm not okay. Εσείς, δεν ξέρω. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι έχουμε κάποιον να μας παρουσιάσει την έκθεση από το EPRS. Αν χρειαστεί θα τους δώσουμε το λόγο. Προτείνω να αρχίσουμε με εσά και βλέπουμε στη συνέχεια στη συζήτηση. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Περί τίνος πρόκειται. Είναι σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την έκθεση ε, για την εφαρμογή του κανονισμού 01-2005 για την προστασία των ε, ζώων κατά τη μεταφορά γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 ε, του κανονισμού. Καθημερινά μαζικά ε, μεταφέρονται ζώα στην Ευρώπη για άλλα κάτω μέλος ή και προς το εξωτερικό για να σπαγούν Με διάφορες συνθήκες που να επικρατούν και ευχαριστώ και ε, την Υπηρεσία Μελετών ε, για την έκθεση που έχει κάνει. Είναι μεικτή η εικόνα, ε, με προόδους βέβαια, αλλά και πολλά προβλήματα και στο μέλλον θα πρέπει επιγόντως να βελτιωθούν. Ήδη το 2012 διατέλεσα σχεώδηση συγγήτρια για μια έκθεση πρωτοβουλία σχετικά με την πρόστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους και για μένα ενδιαφέρον, να μην πω θλιβερό βασικά, ότι έκτοτε δεν έχουν αλλάξει πολλά και σήμερα ε, αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τα ίδια ζητήματα με τότε. Και ακόμα τα ζώα μεταφέρονται πάρα πολύ μακριά για πάρα πολύ χρόνο και όχι πάντα σύμφωνα με την ευημερία και ζωή ανάλογα με το είδος του ζώου. Οι ε, χρόνοι ε, αναμονής ε, στα εξωτερικά σύνορα έχουν μειωθεί ελάχιστα και αν δείτε τον καύσωνα που επικρατούσε φέτος το καλοκαίρι καταλαβαίνετε τα δράματα που ζήσαμε και γενικά ε, τα μέτρα δεν είναι σποραδικά, αποσπασματικά και καθόλου ενία. Ο κανονισμός είναι του 2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Βεβαίως έχει σημαντικές αλλαγές κάνει και βελτιώσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ακόμα και μεγάλα και πολλά. Και κρίμα που σήμερα συζητούμε μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο συνομιλητής αυτό το θέμα κανονικά θα ήταν ε, κατά κύριο λόγο τα κράτη-μέλη. Γιατί τα, προγράμματα, τα προβλήματα μάλλον αυτά, πού οφείλονται, ότι χωλαίνει η ε, εφαρμογή ε, του κανονισμού στα κράτη-μέλη δεν ε, γίνεται πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα και παντού. Και τώρα απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κρίμα που πολλά από τα μέτρα που εσείς έχετε προγραμματίσει έχουν καθυστερήσει μέχρι και πέντε χρόνια και μεταξύ αυτών οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Οι όροι και οι συνθήκες μεταφοράς είναι ενδιαφέροντα για μας στοιχεία όχι μόνο από τη σκοπιά της μεταφοράς των ζώων, αλλά και ως Επιτροπή Περιβάλλοντος που θέλουμε την ενιαία υγεία, την προσέγγιση αυτή που λέγεται One Health, για τη δημόσια υγεία και για να είναι υγιείς οι άνθρωποι και το υγιές το περιβάλλον. Εμείς δεν το βλέπουμε από τη σκοπιά των ζώων αμυγός δηλαδή. Φυσικά Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και ε, στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων. Το στρες και η ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά τους ε, αφορά και τα τρόφιμα. Ε, όταν οι συνθήκες είναι κακές ως προς τον υγιεινή υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης και διάδοσης νοσημάτων. τώρα, για την γνωμοδότηση, μερικά σημεία που προτείνω στο σχέδιο της γνωμοδότησης ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλους περιορισμούς ε, ως προς την έκταση του κειμένου κτλ. Ε, η εφαρμογή είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν είναι αρμόδια περισσότερο του ενός κράτη-μέλη ε, για τις φορτωτικές ας πούμε και τα διάφορα συνοδευτικά όργανα. Ε, θα πρέπει ε, να τηρείται ε, ε, πολύ ο κανονισμός 1 του 2005. Η χρόνη μεταφοράς τώρα. Και αυτό είναι πάγιο αίτημα που το τονίζουμε και πάλι. Για τη σφαγή θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα οκτάωρο μέχρι το σφαγείο. Ε, βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος φόρτωσης. Και ανεξάρτητα αν μεταφορά είναι σε ξηρά ή σε θάλασσα ή σε υδάτινη εδώ. Η καθυστερήση στα σύνορα, πραγματικά λυπηρό. Αυτό προκαλεί στα ζώα ε, πόνους, ε, δεινά και ε, στρες, ε, άγχος. Ε, θα πρέπει να λυθεί αυτό και να βελτιωθεί το συντομότερο από τα κράτη-μέλη. Γενικά γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές ε, βάσει του κανονισμού 1-2005 έχει μειωθεί ο ρυθμός των ελέγχων όμως παρόλο που έχει αυξηθεί ε, ο ρυθμός ε, των μεταφορών ζών των ζώων. Θα πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος για τη μεταφορά ζών των ζώων υπάρχει και ε, ένα θέμα ορισμού για τον κίνδυνο. Δηλαδή υπάρχει το επιχείρημα ότι κάνουμε περισσότερους ελέγχους όταν υπάρχει ρίσκο. Ποιο είναι αυτό το ρίσκο. Τα κράτη-μέλη και οι μεταφορείς θα πρέπει να τηρούν αυστηρά την αντίστοιχη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, πάντα βάσει του κανονισμού 1 του 2005 και καλούμε τα κράτη-μέλη να κάνουν περαιτέρω ελέγχους. Ξέρουμε ότι εδώ Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παραθυράκι ε, για τους χρόνους μεταφοράς ε, μέχρι τα σύνορα, πώς θα ρυθμίζουν τα κράτη έτσι για να παρακάμπτουν ε, κάποιες διαδικασίες και αποφάσεις. Καλούμε ρητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει κίνητρα ε, στους ε, ε, κτηνοτρόφους να σφάζουν τα ζώα τους στο πλησιέστερο σφαγείο για να μην τα πηγαίνουν πολύ μακριά για να σφαγούν. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανατρέξει σε καινοτόμες λύσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να, να εγκρίνονται και να δίνεται άδεια Αξιόπλο σε πλοία ε, που ε, είναι για τη μεταφορά των ζώων όταν αυτά δεν ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Επίσης, οι κυρώσεις ε, και πρόστιμα θα πρέπει να εξομοιωθούν από χώρα σε χώρα γιατί είναι πολύ διαφορετικά και γίνονται και εκεί παρακάμψεις. Υπάρχουν χώρες μέλη που επιβάλλουν πρόστιμα το οποίο αντιστοιχεί σε ένα δέκατο με το πρόστιμο της διπλανής χώρας. Φυσικά έχουμε και άλλα αιτήματα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε αυτές τις λίγες σειρές της νομοδότησης. Θα υπάρξουν λοιπόν συμπληρωματικές τροπολογίες ε, και βεβαίως θα δούμε και την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, για τη μεταφορά των ζώων και την ευημερία τους και θα τα συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές. Χαίρομαι γι' αυτή. Είναι απλώς εντός εισαγωγικών έκθεση πρωτοβουλίας αυτή, αλλά μπορεί να βοηθήσει για να βελτιωθεί ε, η ευζοία των ζώων, αλλά και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντεμισμάκερ, ε, σκιώδη εισηγητή του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάντεμπαχ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Γενικά συμφωνούμε 100% μαζί της. Η ευημερία των ζώων είναι πολύ ψηλά και στις δικές μας προτεραιότητες και ιδιαίτερα η εκτέλεση του κανονισμού για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Αυτό είναι μια παλιά πληγή και καημός και δικός μου. Είχα κάνει και μια γραπτή ερώτηση το 2016 και εξέφρασα την ανησυχία μου ε, για την ευημερία των ζώων όταν εξάγονται ζώντα ζώα προς τις χώρες. Έχουμε και ένα intergroup για την ευημερία των ζώων και επανειλημμένα έχουμε ακούσει εμπειρογνώμονες, έχουμε δει μελέτες σχετικά και επίση ζητούμε να περιοριστεί ο χρόνο μεταφορά σε ένα οκτάωρο. Αυτό το, το κόμμα μου παγίως το έχει στηρίξει και προωθήσει και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί τώρα μια ε, ε νομοδότηση και επαναλαμβάνω καλωσορίζω τη γνωμοδότηση κυρίας Κάτεμπαχ και χαίρομαι για το οκτάωρο που προτείνεται και είναι και προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν και θα το στηρίξουμε απολύτως. Η μοναδική αλλαγή που θα έκανα εγώ σε αυτή την παράγραφο ποια είναι. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα ζώα που προορίζονται για σφαγή, που πάνε στα σφαγεία και τα υπόλοιπα ζώα, που συνήθως πηγαίνουν για εκτροφή. Για ποιο λόγο να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Νομίζω θα ήταν σκοπιμότερο να τα βλέπουμε ενία. Η μελέτη EPRS της Υπηρεσίας Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ε, η εφαρμογή του κανονισμού και μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα και οφείλει να εφαρμόζεται καλύτερα. Το λέει και η δική σας γνωμοδότηση. Θα κάνω μερικές τροπολογίες συμπληρωματικέ. Ε, γενικά συμφωνώ πάρα πολύ με τα όσα λέει η Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάιτεμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα, είναι πιο εύκολο. Ε, καταρχάς, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της γνωμοδότηση. Ε, παρακολούθησα και εγώ τις ε, συζητήσεις στο Intergroup για την ευημερία των ζώων και έχω συζητήσει και με πυρογνώμονες. Έχουμε δει και ντοκιμαντέρ, τα ξέρετε όλοι αυτές τις σκηνέ ε, που μας καλούν σε δράση. Δεν επιτρέπεται να προσπαθούμε παντού και στη γεωργία να ενισχύουμε όσο γίνεται την ευζοία και μετά ξαφνικά στις μεταφορές αυτό να χάνεται να μην ασχολούμαστε. Μερικά σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο γνωμοδότησης και υποστηρίζω απολύτως είναι ε, ο ρυθμός των ελέγχων που έχει μειωθεί ε, το τελευταίο διάστημα από 2,3 εκατομμύρια σε 1,3 εκατομμύρια. Έχουμε χάσει 1 εκατομμύριο ελέγχου. Και πραγματικά χρειάζεται εναρμονισμένο έλεγχο που δεν γίνεται καθόλου κουβέντα γι' αυτό. Επίση θα πρέπει να δούμε και τα πρόστιμα. Στην παράγραφο 9 αναφέρονται αυτά. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι ούτε καν. Ε, μάλλον δεν επιβάλλεται ούτε καν πρόστιμο όταν διαπιστώνεται παράβαση. Επίσης, έχουμε πρόβλημα με τις εξαγωγέ ε, σε τρίτε χώρες, τα είπε και ο κύριος Δεμέσμακερ. Από το 2016 όμως εμείς έχουμε ε, πιστεί στην προσοχή. Έχετε δει τις εικόνες. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Είναι παράδεκτα πράγματα αυτά. Δεν είναι τρόπος μεταχείρισης των ζώων αυτό. Και μάλιστα σε ε, ευρωπαϊκή επικράτεια και μόλι φύγουν από την ευρωπαϊκή επικράτεια επιδεινώνεται η κατάσταση. και οι διάφοροι κτηνίατροι αδιαφορούν, δεν αναλαμβάνουν τη ιδέουσα δράση. Και πραγματικά είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέλνει εκεί καλούς υπαλλήλους και, ε, υπαλλήλους και να γίνονται καλά οι έλεγχοι. Ε, θα κάνω κι εγώ κάποιες τροπολογίες Ξέρω ότι είναι δύσκολη η επιβολή τη νομοθεσία και ακούω από του ενδιαφερόμενου ότι είναι δύσκολο να συνδυαστεί με την ε, νομοθεσία για τι μεταφορέ. Γι' αυτό χρειάζεται μια ενιαία αντιμετώπιση ολιστική όπως τη λέμε τώρα για να μην έχει αρνητική επίδραση η γενική νομοθεσία των μεταφορών στη νομοθεσία για τι μεταφορέ των ζώων. Επίση θα πρέπει να υπάρχουν και χώροι ανάπευση και χώροι συγκέντρωση. Σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχουν αυτοί. Ε, τότε πώς να τηρείς ε, το χρόνο οδήγησης αν δεν μπορείς να σταματήσεις κάπου να ξεκουραστείς. Είναι πάρα πολύ ε, κακές οι συνθήκες. Και εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς ε, θα βελτιώσουμε την νομοθεσία. Και να υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να έχουν χώρους ανάπαυσης. Ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΕ. Ο κύριος Σεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια Κάριν Κάντενμπαχ για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης. Συνάδελφοι, ε, στις θερινές διακοπές ε, Πήγα στην Σλοβενία και την Κροατία για να αποκτήσω εικόνα σχετικά με τις ε, μεταφορές ε, ζώων. Και αυτά που είδα και έζησα εκεί ήταν συγκλονιστικά. Στην Σλοβενία, στο, στο, σε ένα λιμάνι, ήταν και η συνάδελφος Χάζενκαμπ και είδαμε και μάλλον υποστήκαμε ε, δράσεις από πλευράς της αστυνομίας που θέλουν να προστατεύσουν τους μεταφορείς, ε, όχι όμως ε, να διαφλάξουν τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ε, ενώ γνώριζαν ότι είμαστε ευρωβουλευτές, δεν μας σεβάστηκε καθόλου η αστυνομία. Θέλανε να μας απαγορεύσουν ε, να πάρουμε θερμοφωτογραφίες ε, των ε, μεταφορών ζώων και μας απείλησαν. Και 200 ευρώ έπρεπε να πληρώσω στους αστυνομικούς προτού επιστρέψω για να μου δώσουν πίσω το διαβατήριο. Είδαμε θερμοκρασίες ε, πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Ε, σχεδόν 40 ε, βαθμοί ήταν η θερμοκρασία σε κάποια φορτηγά, κανένας όμως δεν παρενέβη. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Και όταν ενημερώσαμε την ιατρική υπηρεσία από το τηλέφωνο, κανείς δεν ήρθε. Και η αστυνομία αρνήθηκε να ελέγξει τα φόρτηγα. Αυτή είναι η προστασία των ζώων στην Ευρώπη και αυτό είναι ντροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει. Μας λέει ψέματα, λέει ψέματα και στους πολίτες, ισχυρίζεται ότι ε, το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών ζώων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και μετά από αυτά στο λιμάνι Κόπα πήγαμε στην Κροατία όπου είδαμε πάλι μεταφορές ζώων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ακόμη και από την Λιθουανία. Και ήταν φρικτά αυτά που είδαμε και φωτογραφίσαμε και ιδιαίτερα αυτά που είδαμε να υφίσταται ένα ζώο το οποίο ε, τραυματισμένο και... Ε, ε, με φωνές ε, μεταφέρθηκε σε ένα πλοίο. Ήταν απίστευτα αυτά που είδαμε. Είναι απίστευτο αυτό να συμβαίνει στην πολιτισμένη Ευρώπη. Και σίγουρα δεν ήταν ε, μεμονωμένο περιστατικό αυτά που είδαμε. Τα... Το φωτογραφικό υλικό ε, που έλαβα θα το στείλω στον Επίτροπο Αντρικάητης. Θα το δείτε και στη γερμανική τηλεόραση και μπορείτε να περιμένετε αντιδράσεις από του ανθρώπους. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ε, πώς πραγματοποιούνται οι μεταφορές ε, στην Ευρώπη και θα πρέπει να σκεφτούν γιατί ακόμη η πλειοψηφία των ε, εκλεγμένων εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ε, ε, κλείνουν τα αυτιά και τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν στις μεταφορές των ζώων. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την κατάσταση αυτή. Και εδώ στο Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει ποτέ να ξαναμιλήσουμε για ηθική εάν δεν κάνουμε κάτι για να δώσουμε τέλος σε, σε αυτήν την ταλαιπωρία των ζώων δεν πιστεύω ότι χρειάζονται τροπολογίες στην έκθεση της συναδέρφου. Ελπίζω να συμβάλλει σε αλλαγή της κατάστασης και προσβλέπω στη συζήτηση με τους άλλους σκιώδεις συζητητές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στο EFDD, στο σκιώδη του EFDD, την κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ε, συνεργάστηκα για αυτή την έκθεση. Ήμουν σκιώδης ε, στην Επιτροπή Αναφορών όπου συντάξαμε μια καλή γνωμοδότηση την οποία ελπίζουμε θα λάβει υπόψη η Επιτροπή Γεωργίας ε, σε όλο το μέγεθος. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή για τη μεταφορά των ζώντων ζώων. Είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων καταγγελιών και αναφορών από Ευρωπαίους πολίτες, ε, πολλές έρευνες, ε, πολλές καταγγελίες από Ευρωπαίους πολίτες και εδώ φυσικά οδηγούμαστε και δεν πρέπει να το, ε, να το ξεχνάμε, οδηγούμαστε σε κάτι τέτοιο από το ότι η διάσκεψη Προεδρών αρνήθηκε να συστήσει μία επιτροπή ερευνητική, εξεταστική επιτροπή που ζητήθηκε από πολλοί αριθμούς ευρωβουλευτές. Δεν είχαμε καν τη δυνατότητα να ψηφίσουμε για τη σύσταση μιας τέτοια ε, εξεταστικής επιτροπής ε, στην Ολομέλεια. Δεν μας δόθηκε καν η δυνατότητα. Αυτό πλήττει τα δικαιώματα και τι ε, δημοκρατικέ αρχές που θα έπρεπε να ισχύουν σε αυτό τον οίκο. Πάμε τώρα ξανά στην έκθεση όμως που συζητάμε σήμερα. Εγώ είμαι ικανοποιημένη από τις προσπάθειες της συναδέλφου Κάντεμπαχ. Αποτελεί εξαιρετική βάση εξαιρετικό εφαλτήριο. Μια έκθεση από την οποία ελπίζω θα μπορέσουμε να μεταπηδήσουμε ε, σε ένα σαφές μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο κανονισμός αυτός έτσι όπως έχει δυστυχώς έχει πολλά κενά όσον αφορά την εφαρμογή του. Θα ήθελα επίσης να είναι σαφές ότι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα για τη μεταφορά εκατομμύριων ζώων, ζώντων στην Ευρώπη είναι ανεπαρκείς. Θα χρειαστεί να καταδικάσουμε καθαρά όσους ε, ε, παραβιάζουν έτσι τα πρότυπα τη ευημερία των ζώων και τη καλή μεταχείριση των ζώων και ειδικότερα του ελεγκτικού οργανισμού που σήμερα νύπτουν τα σχήρα του. Ουσιαστικά δεν του ενδιαφέρει καθόλου σε τι συνθήκε ε, υποχρεούνται να ταξιδεύουν τα ζώα. Το έχουμε υπενθυμίσει, το επαναλαμβάνω και εγώ. Πολύ μεγάλε αποστάσει, υψηλέ θερμοκρασίε, υψηλότατε θερμοκρασίε σε απαράδεκτα επίπεδα, στέρηση από νερό, ε, τροφή. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα προβλήματα τα οποία τακτικά, τακτικά ε, ε, μα καταγγέλουν διάφοροι καταγγέλλοντες, ε, οι οποίοι καταγγέλουν και την απόλυτη απουσία ελέγχων μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης και Τουρκίας ε, λείπουν τέτοια έλεγχη, αλλά όχι μόνο. Είναι μια τεράστια απάτη αυτή η έλεγχη. Όσοι ζουν την πραγματική κατάσταση μας λένε ότι δεν, δεν υπάρχουν τέτοια έλεγχοι. Ο Επίτροπος Ανδριουκάητης μας απάντησε σε μια επιστολή που στείλαμε πριν κάποιο καιρό και μας μίλησε για compliance 100%, συμμόρφωση 100%, παράδεκτη απάντηση κατά την απόψή μου. Οπότε επαναλαμβάνω αυτό το σχέδιο Έκθεση αποτελεί εξαιρετική αφετηρία. Συμφωνώ στα σημεία που επισημάνθηκαν. Να επαναλάβω κάποια που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να βαθύνουμε λίγο παραπάνω ή να συμπληρώσουμε ε, στην έκθεση αυτή. Ε, για παράδειγμα, η μη τήρηση των ε, περιόδων διαλύματος, ο υπερπληθυσμός, η έλλειψη νερού, οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες Όλες αυτές οι πτυχές θα μπορούσαν να αναφέρονται πιο λεπτομερώς εντός της έκθεσης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο στην εξαιρετική δουλειά που έχει ήδη γίνει. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε τώρα σε επιπλέον σχόλια από τα μέλη των Επιτροπών. Η κυρία Μέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ ιδιαίτερα την κυρία Κάντεμπαχ για την έκθεση αυτή. Αρμόδια επί της ουσίας ε, επιτροπή που καταρτίζει την έκθεση είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Και εμείς θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Ε, είδαμε ξεκάθαρα ότι έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος μπορεί να είναι καλογραμμένος, αλλά στην ε, υλοποίηση αφήνει τόσα παραθυράκια που τελικά δεν μας βοηθάει καθόλου να βελτιώσουμε την προστασία των ζώων. Αρκετά παραμείναμε θεατές. Επανειλημμένα ε, προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν. Η χρόνη αναμονή στα εξωτερικά σύνορα είναι τεράστια, καθώς επίσης και ε, ε, οι ε, ρυθμίσεις για, τις, ε, για τους χώρους συγκέντρωσης. Ξέρουμε ότι εκτός της Ένωσης σε καμία περίπτωση τα, τα ζώα αυτά δεν εκφορτώνονται για να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό. Και τα προβλήματα είναι και στη μεταφορά των, των μόσχων αλλά και των μικρών θηλαστικών. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε και να φροντίσουμε να τηρείται το οκτάωρο στις μεταφορές και αυτό δεν έχει να κάνει είναι προσωπική μου πεποίθηση κιόλα ότι ε, όχι μόνο το οφείλουμε στα ζώα, γιατί εγώ είμαι αγρότησα και κτηνοτρόφος και πολύ υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη ε, και ακριβώς όπως προσέχω τα ζώα μου στην εκτροφή θέλω να είναι προσεγμένα και στις μεταφορές. Επίσης υπάρχουν και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μακρινές Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ε, έχουν συνειδητοποιηθεί ε, και μας δείχνουν το δρόμο, δεν μεταφέρουν πια ζωντανά εγωπρόβατα. Ε, in ordnung, aber λοιπόν, οι κανονισμοί μπορεί να είναι εντάξει, αλλά δεν εφαρμόζονται σωστά. Και εγώ ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει εάν σκέφτεται να μειώσει τις μεταφορές ζώων προσφαγής σε τρίτες χώρες, απάντηση όχι η απάντηση ήταν ότι έχουμε ένα εμπόριο που βασίζεται σε αξίες. Χαιρετίσματα. Αξίες δεν είναι και η προστασία των ζώων. Ε, θα πρέπει να επιδείξουμε ε, θάρρος και να πούμε ότι απαγορεύουμε τις μεταφορές και τις εξαγωγές ζώων των ζώων εκτός της Ένωσης προσφαγή. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Είμαι πεπισμένη ότι όταν έχουμε ε, ζώα παραγωγικά που σφάζονται κοντά στην εκτροφή, η ποιότητα του κρέατος είναι πολύ καλύτερη παρά να ε, διανύουν τέτοιες αποστάσεις τα ζώα και να στρεσάρονται με αυτόν τον τρόπο. Ε, λοιπόν, μετά από όσα μας είπε ο συνάδελφος ΕΚ, ε, είδαμε ότι και εντός της Ευρώπης δεν είναι όλα καλώς και για μένα το να μεταφέρονται ζώντα ζώα με πλοία είναι απαράδεκτο και αφόρητο πλέον. Ε, αν ε, ε, έχουμε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και αντίστοιχες κυρώσεις και πρόστιμα, να το σκεφτούμε. Τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε για τους στόχους μείωσης καυσαερίων και εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα από τα φορτηγά. Και επιβάλλονται ε, τεράστια πρόστιμα ε, στα φορτηγά ε, όταν εκπέμπουν έστω και ένα γραμμάριο περισσότερο από το κανονικό. Για τις μεταφορές των ζώων του ζώων τι θα κάνουμε. Τα παραγωγικά ζώα που μεταφέρονται εκτός της Ευρώπης χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία αλλά όλα τα υπόλοιπα τα ζώα προσφαγή να σφάζονται στην Ευρώπη. Τα, τα άλλα τα που είναι η προσεκτροφή και εξάγονται προφανώς να εξακολουθήσουν να εξάγονται. Ευχαριστώ και με ενημερώσαν ότι έχουμε αντικαταστάτη του σκιώδου ή των πρασίνων ε, και δίνω το λόγο στην κυρία Μέτς. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους του Keith Taylor και ε, χρησιμοποιώ το κινητό μου τηλέφωνο ε, για να σας παρουσιάσω τις παρατηρήσεις του και συμμερίζομαι τις θέσεις του. Οι μεταφορές ζών δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται καθόλου. Ε, εγώ θέλω να έχουμε ομαλό εμπόριο ζώντων ζών και Θέλουμε να προστατεύσουμε εκατομμύρια ζώων από αυτήν την περιττή ταλαιπωρία, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να μειώσουμε και τις μεταφορές και έτσι να έχουμε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ε, μείωση των, ε, και μείωση των εκπομπών. Συμφωνώ με την έκκληση της εισηγήτριας ε, για απαγόρευση όλων των μεταφορών άνω των 8 ώρων. Εγώ θα υποβάλω τροπολογία για να μειώσουμε το όριο αυτό στις 4 ώρες. Και χαίρομαι που η συγγήτρια συμφωνεί με την Ένωση Εκτινιάδρων της Ευρώπης και άλλους που πιστεύουν ότι ε, τα ζώα θα πρέπει ε, να εκτρέφονται και να ε, σφάζονται στις, στην ίδια περιοχή αντί να μεταφέρονται μακριά. Και για να το διασφαλίσουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε περιφερειακά σφαγεία καθώς και κινητά σφαγεία. Επίσης, Συμφωνώ όσον αφορά την ταλαιπωρία των ζώων ε, λόγω της ε, αναμονής στα σύνορα, όπως είναι τα σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Τουρκίας. Πολύ συχνά πρέπει να περιμένουν εκεί μέρες σε, σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ε, έχουμε την ε, απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι οι μεταφορείς ε, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσει του κανονισμού μέχρι τον τελικό προορισμό, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι κακές συνθήκες και η έλλειψη εγκαταστάσεων στα σύνορα τρίτων χωρών σημαίνουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πράξη και γι' αυτό σας καλώ να, καλέσω, να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε μεταφορά ζών των ζώων ε, ε, για σφαγή και επίσης ε, βλέπουμε μεγάλη ε, έλλειψη συμμόρφωσης ε, σε ευρωπαϊκές χώρες. Θέλουμε λοιπόν μια σειρά μέτρων όπως είναι τα καλύτερα πρότυπα οχημάτων, περισσότερη κτηνιατρική έλεγχη και μαύρη λίστα των οικονομικών φορέων που να καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης οι κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό εφαρμογής που τους παρέχεται στο πλαίσιο του κανονισμού. Ε, θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που ήδη έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάθε χρόνο πάνω από 4 εκατομμύρια βοηθοί, εκατομμύρια ε, άλλων ειδών, ε, ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη και πολύ μακριά στο εξωτερικό. Γουρούνια, πουλερικά, άλογα κτλ. Ε, είδα ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για το πώς ε, μεταφέρονται ζωά από τα ευρωπαϊκά λιμάνια με πλοία. Και αυτά που είδα ήταν τόσο φρικτά που ε, απευθύνθηκα ε, σε κάποιες οργανώσεις προστασίας των ζώων. Όλα αυτά ήταν τη δεκαετία του 80 και τώρα 30 χρόνια αργότερα δεν έχει αλλάξει τίποτα πραγματικά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχουμε περίπου 100% συμμόρφωση. Μα τι είναι αυτό, δεν ισχύει καθόλου. Φέτος το καλοκαίρι πήγαμε το συνάδελφο ΕΚ και μετά από το συνάδελφο Τόματς Βάιτσαλ στη Σλοβάνια. Ε, Σλοβενία και στην Κροατία, σε δύο λιμάνια, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, για να δω πώς εξάγονται τα ζώα. Και αυτά που είδα πραγματικά δεν περιγράφονται. Όλα τα φορτικά που έφταναν εκεί για να φορτώσουν τα ζώα, ε, είχαν μοσχάρια φορτίο και όλα τα φορτηγά που έφταναν εκεί ήταν παράνομα ε, με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν τηρούσαν την νομοθεσία και δεν έτρεχε τίποτα. Ε, μετρήσαμε τη θερμοκρασία ε, το πρωί και ήταν πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Και σε όλα τα φορτηγά ήταν υπερβολική θερμοκρασία. Τα ζώα ήταν βρώμικα, ήταν χάλια και περίπου θερμόπληκτα απόντες οι εκτινίατροι και καμία διαχείριση. Η αστυνομία ήθελε να προστατεύσει τη βιομηχανία, τον κλάδο και να απαγορεύσει σε εμά να φτάσουμε στα ζώα. Αυτή ήταν η δουλειά της αστυνομίας. Ε, θέλησαν να μας εκφοβήσουν και μάλιστα ήταν και θέμα, εκτός από ε, εκφοβισμό, και θέμα διαφθοράς και το λέω το λέμε στην έκθεση ότι υπάρχουν προβλήματα, όλο και περισσότερες μεταφορές, λιγότερη έλεγχη, η χρόνη μεταφοράς είναι πολύ μεγάλη, χρόνη αναμονής ε, στα σύνορα επίσης και δίνονται άδειε που κανονικά δεν θα έπρεπε να δίνονται. Και δεν μιλάω μόνο για τις μεταφορές διαθαλάσσεις. Φανταστείτε ένα ζώο που φεύγει από την Ιρλανδία από μια εκτροφή, μπαίνει σε ένα φορτηγό και πάει στο λιμάνι και μετά μπαίνει σε ένα πλοίο και φτάνει σε ένα άλλο λιμάνι. Μετά μπαίνει σε άλλο φορτηγό, διασχίζει όλη την Ευρώπη μέχρι το λιμάνι Κόπερ στη Σλοβενία. Μετά το ξεφορτώνουν, το βάζουν σε άλλο πλοίο και πάει στο Λίβανο, ξέρω εγώ, ή στο Ισραήλ για να σφαγεί. Και όταν φτάνει εκεί, άντε πάλι φορτηγό για να πάει στον τελικό του προορισμό. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι Εντάξει, η συμμόρφωση πάει καλά. 100% σχεδόν και δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν ισχύει αυτό. Ε, η κατάσταση είναι φρικτή και απέσια και δεν μπορεί ούτε να απαντά αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε να συμπεριφερόμαστε έτσι στα ζώα. Επανέρχομαι στη γνωμοδότηση. Όπως και στην ε, μελέτη IPRS, η εστίαση είναι πάρα πολύ στα ζώα φαγή και όχι στα ζώα προς εκτροφή. Τα είπε και ο συνάδελφος Ντεμέσμακερ και υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ κατά την άποψή μου. Ας πούμε, στα ζώα ε, που πηγαίνουν για εκτροφή υπάρχουν έγκυες αγελάδες ή ε, ε, μικρά μοσχάρια. Ακόμα θυλάζοντα που δεν έχουν απογαλακτιστεί. Εδώ δεν έχουν ούτε νερό στα φορτηγά πολλές φορές. θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τα ζώα αυτά. Και χρειάζεται λύση. Λιγότερη περισσότερη έλεγχη, λιγότερες μεταφορές, ε, απαγόρευση εξαγωγών, ε, κοντινά ασφαγεία. Όλα αυτά είναι μέτρα που προτείνονται, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως σύστημα εκτροφών ε, και γεωργίας και παραγωγής τροφίμων με περισσότερα φυτικής προέλευσης τρόφιμα και λιγότερα ζωικής προέλευσης. Και τέλος, Πρόεδρε, πέρυσι 220 βουλευτές, δεξιοί ή αριστεροί από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ζητήσαμε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Μεταφορές των Ζώων. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν μια αρχή, αλλά δεν πρόκειται και η έκθεση να οδηγήσει πουθενά, γιατί ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον, η Κομισιόν μας παραπέμπει στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν, θα πρέπει να γίνει κάτι πιο ριζικό. Και επιμένουμε πάρα πολύ στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και ελπίζω οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος να ακολουθήσουν την σύστασή μου αυτή. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Να, σας, να κάνω και εγώ μια προσωπική παρατήρηση ως ε, Ευρωβουλευτής, όχι ως Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και τους κοιόδης ε, και ο Σλοβαίνος φυσικά κάνω τις παρατηρήσεις αυτές. Ε, η μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι φρικτό και έχουμε και φρικτά σφαγεία σε κάποια μέρη έξω από τα σύνορά μας. Ρόλος μας λοιπόν, ρόλος συγγνώμη πολλών είναι περισσότερο να, το, να κρύβουν το πρόβλημα παρά να το λύνουν. Ελπίζω λοιπόν η συζήτηση αυτή και οι περαιτέρω δραστηριότητε ε, των ενδιαφερομένων να συμβάλλουν σε καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού αλλά και για τη δημιουργία νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των ζώων. Τέλος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκούτελα και μετά θα πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Κάρεν Κάντεμπαχ. Ήταν εξαιρετική η έκθεση αυτή. Έχω τα ίδια συναισθήματα με σας κύριε Πρόεδρε. Ανησυχώ. Αλλά παίρνω και κουράγιο ακούω τους συναδέλφους που ανησυχούν για τη σημερινή κατάσταση. Όταν δεν υπάρχει νομοθεσία, αισθάνεται κανείς ε, ανήσυχος. Αλλά όταν υπάρχει νομοθεσία η οποία όμως δεν τηρείται, η ενόχληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι ε, κάπως ηρωνικό. Αν δεν είναι επαρκώς δυνατή η νομοθεσία και όταν δεν την τηρεί ο κόσμος, αποτελεί τροχοπέδι για την πρόοδο στην ουσία. Μίλησαν συνάδελφοι για το πόσο άσχημο είναι να παλεύει κανείς για 30 χρόνια, να πετυχαίνει την νομοθεσία και τελικά η κατάσταση για το ζώο να μην αλλάζει. Παίρνω κουράγιο λοιπόν ακούγοντάς σας συνάδελφοι να εκφράσετε όλες αυτές τις ανησυχίες ε, ε, που βλέπετε ζώα τα οποία είναι ε, ζώα με συναισθήματα, είναι όντα με συναισθήματα και να τα βλέπει κανείς να υποφέρουν από τη ζέστη, από την έλλειψη νερού, από τις αρρώστιες κατά τη μεταφορά μιλάμε για νεαρά ζώα που χρειάζονται τις μητέρες τους και θυμώνω πραγματικά πολύ όταν βλέπω την κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη και νομίζω ότι εδώ έχουμε και τους πολίτες με το πλευρό μας στο πλευρό μας σε πολλά κράτη-μέλη πολλοί κόσμος θεωρεί ότι δεν έχουν γίνει αρκετά πολλοί κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η νομοθεσία έτσι ακριβώς όπως το παρουσιάζει η Κάραν σήμερα Πολλοί κόσμοι θέλουν να υποστηρίξει πιο αυστηρά ε, μέτρα ώστε να μην συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Συναισθηματικά ε, αισθάνομαι μεγάλη φόρτιση, αλλά χαίρομαι που ακούω και του συναδέλφου που θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση. σα. ευχαριστούμε λοιπόν Κάρεν και όλους σας. Ευχαριστούμε. Δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άννα Ραμιρεσέλα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή. Η Κομισιόν θεωρώ ότι είναι εξαιρετική, πολύ καλή αφετηρία και πολύ ισορροπημένη. Θα το έχετε ξανακούσει, η μεταφορά των ζώων αποτελεί προτεραιότητα ε, τη Κομισιόν στα θέματα ευημερία των ζώων και καλής μεταχείριση των ζώων. Το μελετάμε και αναγνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σημειώνεται κάποια βελτίωση και εμείς πιστεύουμε ακραδάντα στην Κομισιόν ότι η κατάσταση δεν είναι καλή γενικά, αλλά υπήρξαν μεγάλες βελτιώσεις. Κάποια πράγματα έχουν γίνει σωστά και κάποια άλλα δεν έχουν γίνει σωστά. Ε, και όταν ο κανονισμός θα εφαρμοστεί όπως πρέπει, θα παρέχει την επαρκή προστασία στα ζώα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχουμε πολλά μέτωπα στην Κομισιόν αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη και με άλλους ενδιαφερομένους όπως ΜΚΟ, ε, και διάφορους φορείς ε, για να προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα που παρουσιάσατε και εδώ όσον αφορά τις εξαγωγές των ζώων, τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη ε, τόσο στην πλατφόρμα όσο και στο δίκτυο των σημείων επαφής. αναμένουμε την τελική έκθεση, την, τελευταία έκδοχη της έκθεσης από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάρεν, δεν ξέρω αν θέλετε να αντιδράσετε, να απαντήσετε στην Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες στον τομέα αυτών. Και εμείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να στραφούμε και προς τα κράτη-μέλη. Άλλωστε έχουμε και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το θέμα των μεταφορών, αλλά... Συγγνώμη, το, την απόφαση του δικαστηρίου, ε, που ε, δείχνει ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα των μεταφορών, είναι γενικά το πρόβλημα πώς ε, αντιμετωπίζουμε τα ζώα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για την συνεισφορά τους, κοιτώ και την Γιούτε. Ναι, καταλαβαίνω την δυσαρέσκεια όταν βλέπουμε την κατάσταση επιτόπου. Απ' την άλλη νιώθω αισιόδοξη όταν ακούω τις απόψεις των συναδέλφων. Πιστεύω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Όπως ε, και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα, είμαι αναπληρωματικό μέλος ε, της Επιτροπής ε, Γεωργίας και θα καταβάλω προσπάθειες ώστε να φροντίσουμε τα δικά μας συμπεράσματα να περάσουν στην τελική έκθεση. Προσλέπω στην καλή συνεργασία. Πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια Ευρώπη που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ευημερία των ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 14 Νοεμβρίου στις 11, ψηφοφορία στην ΕΝΒΙ 6 Δεκεμβρίου και ψηφοφορία στην Άγκρη 21 Ιανουαρίου. 14 ε, η προθεσμία κατάσταση ε, τροπολογιών. Ναι, πράγματι. Α, συγγνώμη, λέει κυρία Κάντενπαχ, νόμιζα ότι είπατε 18. Όχι, πράγματι, 14 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και περνάμε στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις. Ε, πρόταση ψηφίσματος. Πρώτα, θέλω να δώσω το λόγο στους συνεισήγητες. Καταρχάς, στην κυρία Σάλντε Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πιατικάινεν βρίσκεται στο Ελσίνκι σήμερα για την ε, διάσκεψη του ΕΛΚ. Ε, αυτό πάντως που θέλουμε με το ψήφισμα και με την προφορική μας ερώτηση είναι να ε, καλέσουμε ε, όλους για υποστήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Έτος για πιο πράσινες πόλεις ε, το 2020. Θα είναι πολύ χρήσιμο να εστιάσουμε στο πώς μπορούν να γίνουν πιο πράσινες οι πόλεις μας. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε πιο πράσινες πόλεις, διότι αυτό θα είναι καλό για το περιβάλλον και καλό όσον αφορά την προστασία του κλίματος. Με πιο πράσινες πόλεις θα ενισχύσουμε την βιοπικιλότητα, θα μειώσουμε τα υγρά απόβλητα κλπ. Επίσης θα έχουμε καλύτερα ε, συστήματα απορροής των ε, νερών ε, της βροχής και επίσης μπορούμε να δεσμεύσουμε διοξίδιο του άνθρακα με πιο πολλά δέντρα για παράδειγμα και μπορούμε να μειώσουμε και την κατανάλωση θέρμανσης και ενέργειας στα κτίρια. Έχει λοιπόν να κάνει το θέμα αυτό με την αλλαγή του κλίματος. Επίσης, θα έχει θετικές επιπτώσεις για την υγεία. Εάν ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πόλεις, μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα θορύβου που αποτελεί πρόβλημα για πολλούς πολίτες. Μπορούμε να μειώσουμε και την ρήπανση του αέρα. Από όλες τις απόψεις ε, λοιπόν ε, θα είναι χρήσιμο να υποστηρίξουμε τις πόλεις μας και να τις βοηθήσουμε να γίνουν πιο πράσινες. Πιστεύουμε ότι ένα ευρωπαϊκό έτος για πιο πράσινες πόλεις ε, θα μας βοηθήσει να εστιάσουμε στο θέμα αυτό, να δώσουμε περισσότερη ορατότητα στο θέμα αυτό και να μάθουμε ένας από τον άλλον. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι στον τομέα αυτόν, διότι πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή ε, καλών ιδεών και βέλτιστων πρακτικών ε, είναι καλή μέθοδος ώστε να πετύχουμε κάτι στον τομέα αυτό, να μην χρειάζεται όλοι να επανεφεύρουμε τον τροχό. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες πέρα από την απλή υποστήριξη. Να έχουμε λοιπόν ένα έτος για πιο πράσινες πόλεις στην Ευρώπη, αλλά να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο για ανταλλαγή εμπειριών, ώστε όλες οι πόλεις μας να καταβάλουν προσπάθειες να γίνουν πιο πράσινες. Γι' αυτό έχουμε εκπονήσει το ψήφισμα αυτό. Ε, οι σοσιαλδημοκράτες το στηρίζουμε, διότι είναι καλό για το περιβάλλον, για την υγεία, για το κλίμα και και συνολικά μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών μα. Ε, στηρίζουμε λοιπόν την πρόταση αυτή και ελπίζουμε να υπάρξει ευρία υποστήριξη για το ψήφισμά μα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία και είναι η επόμενη ομιλήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Θεωρώ ότι αυτή η ιδέα με τις πράσινες πόλεις ε, είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. 72% των πολιτών ζουν σε πόλεις και θεωρώ ότι αυτή η ιδέα των πράσινων πόλεων έχει νόημα για, συνδυάζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και βοηθά ε, να ζει κανείς πιο άνετα στις πόλεις. Θα πρέπει να λάβουμε διάφορες πτυχές υπόψη, οικονομικές, κοινωνικές και φυσικά και τις πολιτιστικές. Όλες αυτές εξαρτώνται η μία από την άλλη. Και πρέπει να... Ε, αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη θα μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζωογόνηση των πόλεων και που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να χρησιμοποιηθούν επαρκώς και χωρίς αποκλεισμούς. Ο αγώνας για τις πρασινότερες πόλεις ε, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανεξαρτήτω ε, πόλεων, αλλά με διάφορου τρόπου ανάλογα με την πόλη. Στην Πολωνία, να σα πω τι κάνουμε. Στην Πολωνία τα πράγματα έχουν ω εξή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα προτεραιότητας που εφαρμόζουμε για καθαρότερο αέρα. 24 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ε, ε, έχουν αφιερωθεί σε αυτό και το συνολικό κόστος είναι πάνω από 30 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ε, και οι προσπάθειες λιγότερων εκπομπών είναι οι στόχοι η τηλεθέρμανση επίσης, όλα αυτά θα βοηθήσουν ε, στη μείωση των εκπομπών. Θέλουμε οι πόλεις να μην πνίγονται να μην πνίγονται ε, από τα καυσαέρια και να τηρούμε και τους ε, κανόνες των Παρισίων. Σας ευχαριστώ όλους που υποστήριξατε εδώ την τροπολογία μου. έχουμε μπορέσει να ε, ε, υπογραμμίσουμε εδώ πέρα την τηλεθέρμανση, πράγματι την αστική τηλεθέρμανση στην ε, διότι στην Πολωνία για να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές καυσαερίων πρέπει να αντιμετωπίσουμε το smog, την ατμοσφαιρική ρήπανση και η τηλεθέρμανση αυτή, η αστική θέρμανση θα μπορέσει να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. From the Κυρία Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος. Και καλωσορίζω την πρωτοβουλία αυτού, για αυτό το έτος ε, πιο πρασινών πόλεων. Έτσι θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τι ε, παλιότερε εμπειρίε και πρακτικέ στην Ευρώπη. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίω ζουν σε πόλει. Και οι περισσότεροι πόροι ε, του πλανήτη χρησιμοποιούνται επίση ε, στι πόλει. Ο τρόπος οργάνωσης λοιπόν των πόλεων αποτελεί επίκεντρο της προσπαθειάς μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι πολίτες ε, για βιώσιμη διαβίωση στους πολίτες ε, ε, για αποτελεσματική ανακύκλωση, για αθλητισμό, για ελαχιστοποίηση της χρήσης του αυτοκινήτου, για έξυπνο αστικό σχεδιασμό και για υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι ευκαιρίες που παρέχονται στις πόλεις ώστε να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές που παράγουν οι κοινωνίες μας. Για άλλη μια φορά ανακαλύπτουμε μια αρχαία αλήθεια. Το να περνά κανεί χρόνο σε πράσινους χώρους και σε πράσινες υποδομές έχει πολύ θετικέ επιπτώσει για την υγεία, όπω υπόθηκε και προηγουμένω. Γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται να προωθούμε τέτοιου χώρου πράσινου, όλο και περισσότερο στο αστικό περιβάλλον επίση. Το πράσινο μας προστατεύει από την ακραία ζέστη που συχνά αποτελεί πρόβλημα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις. Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα ε, που έχουν οι πιο πράσινες πόλεις είναι ότι ε, ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερη άσκηση, να αθλητισμό και αυτό βοηθά την υγεία. Σε μεγαλοπόλεις όπως η Βαρκελόνη ή σε κομοπόλεις όπως η πόλη του Λάχτη στη Φιλανδία, ε, σε όλες αυτές τις πόλεις παρατηρούνται πρωτοβουλίες ολιστικής μεταμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει κάποιο φόρουμ αναθεώρησης όλων αυτών των πρωτοβουλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο κύριος Έκχαρτ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ επικροτώ την πρωτοβουλία αυτή. με το Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις, οι πόλεις μας ε, μπορούν να ε, αποτελέσουν ε, υπόδειγμα καλύτερων πόλεων και έτσι να έχουμε βιώσιμες λύσεις για τα προβλήματα του πολιτισμού. Οι πόλεις θα πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένες ώστε να επιτρέπουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και για να μπορούν να αντιδρούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Με πιο πράσινες πόλεις θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Πιο φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν ε, χρήσιμο εργαλείο. Μπορούμε έτσι να επηρεάσουμε την αλυσίδα αξίας ε, για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα. Η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων στις πόλεις ε, συχνά δημιουργούν προβλήματα για το περιβάλλον ε, απέναντι στα οποία δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας. Και γι' αυτό ελπίζω όσοι λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την νέα αυτή πρωτοβουλία να καθοδηγήσουν τους ε, ανθρώπους ώστε να ε, έχουν ε, μεγαλύτερη συνείδηση των θεμάτων βιωσιμότητας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την παρεξήγηση. Ο κύριος Εκ από την ΚΟΕ. Τώρα περνάμε στους πρασίνους. ο κύριος Έκχαουτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ναι, εντάξει, Εκ, Έκχαουτ μοιάζουν τα ονόματα. Ποια η διαφορά, το χάουτι είναι που κάνει τη διαφορά. Θα ήθελα να ε, σας συγχαρώ για το ψήφισμα αυτό. Όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι βλέπουμε να συμβαίνουν όλο και περισσότερα εντός των πόλεων. Και όχι μόνο στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου γνωρίζουμε ότι η κεντρική κυβέρνηση εγκαταλείπει τη συνθήκη του Παρισιού, ταυτόχρονα βλέπουμε ε, πολλές πόλεις να αναλαμβάνουν ε, δράσεις για το κλίμα. Έχουμε τον όλο συνασπισμό που ε, επιμένει στην συνθήκη και βλέπουμε να παρουσιάζει και αποτελέσματα όσον αφορά τις μειώσεις που πρέπει να, βρεθούν, να πραγματοποιηθούν. Βλέπουμε και στην Ευρώπη τις πόλεις να βρίσκουν όλο και πιο βιώσιμους τρόπους. Ε, στις πόλεις λοιπόν βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό το 2020 να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις πιο πράσινες πόλεις και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ε, στην παρουσίαση αποτελεσμάτων, όπου συχνά εμείς στο πολιτικό επίπεδο εδώ στην Ευρώπη αποτυγχάνουμε. Για παράδειγμα, να έχουμε πιο καθαρά αυτοκίνητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφήσαμε στις πόλεις όλες ε, τις ε, δραστηριότητες που πρέπει να αναλυφθούν. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε με καλύτερο τρόπο να υποστηρίξουμε τις πράσινες πόλεις. Χαίρομαι όμως που έχουμε τις πιο πράσινες πόλεις και πολύ ευχαριστώ θα στηρίξω το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο EFDD. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ υποστηρίζω εξ ολοκλήρου το ψηφίσμα αυτό. Θεωρώ ότι οι πράσινες πόλεις είναι ένα σημαντικό θέμα για το μέλλον που μας περιμένει. Η φροντίδα των πολεών μας είναι σημαντική. Πρέπει να είναι όλο και πιο καθαρότερες, να βασίζονται σε πράσινες υποδομές. Ε, έπρεπε είναι, να είναι και ε, κανόνας αυτό εδώ και καιρό. Δεκαετίες όμως κακοδιαχείριση σε πολλές πόλεις της Ευρώπης ε, δημιούργησαν ευάλωτες συνθήκες που διαλύουν τις πόλεις ε, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές ε, κλιματικές ε, καταστάσεις και περιπτώσεις που είδαμε να διατρέχουν την Ιταλία από το βορρά μέχρι το νότο τις τελευταίες εβδομάδες και που γίνονται όλο και πιο έντονες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ε, απερίμωση και νεκρή είναι το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί όλοι αυτοί αν είχαμε φροντίσει περισσότερο τη φύση, αν είχαμε αγαπήσει περισσότερο τον πολιτισμό μα την κληρονομιά μα και είχαμε διατηρήσει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ αστικού ιστού και προστασία του περιβάλλοντο. Γι' αυτό το λόγο η λέξη αντοχή και η αντοχή ω έννοια στι πόλει ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αναλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε αυτό το ψήφισμα μα δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και εγώ συμφωνώ θα πρέπει να αναπτύξουμε τις πράσινες υποδομές για να ενδυναμώσουμε τα θεμέλια των πολεών μας. Συμφωνώ λοιπόν η πρόταση αυτή του να ορίσουμε το 2020 να το ανακηρύξουμε ως έτος των πιο καθαρών πόλεων και η πρόταση του να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης για πιο πράσινες πόλεις μέχρι το 2030 είναι σημαντικό. Είναι θετικό που στρέφουμε την προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση ώστε οι πόλεις μέσα στην επόμενη δεκαετία να κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβάλλουν και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διότι δυστυχώ ε, το βλέπουμε στην πράξη ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά συμφωνώ και με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι πολύ συχνά, σε τοπικό επίπεδο οι δήμαρχοι είναι μόνοι τους ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των θεόρατων προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Ε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε λοιπόν με μεγαλύτερη, πιο στεναρά, συγγνώμη, θα χρειαστεί παρά τη δική μας συμβολή και μια, ένας αστικός προγραμματισμός με ενεργό συμμετοχή των πολιτών μακροχρόνια. Εκεί ακριβώς στα θέματα που θέλουν ε, οι κάθε, ο κάθε Δήμος ξεχωριστά εγώ ως ε, Ιταλίδα πολίτης από τη Λομβαρδία ξέρω ότι οι πόλεις μπορούν να κάνουν περισσότερα ώστε να ξεπεραστεί αυτό το παράλογο ε, αστικό περιβάλλον έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζοντας το περιβάλλον. Πρόσφατα είχαμε μία έκθεση της ΙΣΠΡΑ το 2018 για τη χρήση της γης και η εδαφοκάλυψη στην Ιταλία ε, μειώνεται κατά δύο τετραγωνικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Στη Λομβαρδία είμαστε οι χειρότεροι όσον αφορά τη χρήση αυτή του γεών ε, την καταστροφή των γεών έχουμε φτάσει στο 52%. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Αν συνεχίσουμε έτσι θα επιδεινώνεται διαρκώ η κατάσταση ε, υποβάθμισης του υδρολογικού ε, της υδρολογικής κατάστασης και θα απομακρυνόμαστε από τους στόχους της βιώσιμη ανάπτυξης, ειδικότερα από τον στόχο 15 για τη βιώσιμη χρήση των γεών. Εμεί θα συμβάλλουμε στην εκτίση αυτή με σημαντικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κλείνει ο γύρος των συνεισηγητών, αλλά έχουν ζητήσει και άλλα μέλη το λόγο. Ε, πρώτος ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές αυτού του ψηφίσματος που ανακηρύσσει το 2020 ως το έτος των πιο πράσινων πόλεμων. Ξέρουμε πόσο Μεγάλες είναι οι δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πόλεις μας, η κακή ποιότητα του αέρα, ε, τα κυκλοφοριακά προβλήματα στα ιστορικά κέντρα, τα ακίνητα, ε, οι διάφορες καταστροφές, οι όλο και μεγαλύτερες και ακραίες καταιγίδε. Ε, συμφωνώ λοιπόν με αυτή την πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε τους πολίτες να μεταβούν σε ένα νέο αστικό μοντέλο και καλό την ε, Κομισιόν να παρέσχει επαρκή χρηματοδότηση για την ε, αναδιοργάνωση του αστικού περιβάλλοντος. Πρέπει να πούμε ότι η, αρμονική ανάπτυξη των πόλεων βοηθά και τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, διότι επανεξισορροπείται ε, η επικράτεια σε κάθε χώρα. Η Λισαβόνα θα είναι πράσινη πρωτεύουσα έχει δοθεί το βραβείο μετά χάρη σε πολλές πρωτοβουλίες που έγιναν για την κινητικότητα, για την κοινή χρήση οχημάτων, για, την, για τον καθαρισμό του ποταμού, για τη βελτίωση των συγκοινωνιών και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ε, των δημοσίων κτίριων με περηφάνεια. Ε, βλέπω λοιπόν τη Λισαβόνα να ανακηρύσσεται Ευρωπαϊκή Πράσινη Πόλη του 2020. Στο πλαίσιο αυτού του έτους πιο πρασινών πόλεμων αυτή η πρακτική θα πρέπει να γίνει πιο κοινή ε, ώστε οι πόλεις μας να γίνουν πιο ευχάριστες, ε, ο κόσμος να ζει σε αυτέ. τόσο ευχάριστα όσο και όταν τι επισκέπτεται. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το ψήφισμα είναι μια καλή βάση, καλή αφετηρία παρότι έχουν ακόμα να γίνουν πολλά. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Yes, thank you very much for, um, for the Ευχαριστώ πάρα πολύ μου δίνετε το λόγο και για το ψήφισμα αυτό. Φυσικά η Κομισιόν καλωσορίζει ε, την ναι, προσοχή που δίνει το Κοινοβούλιο στην τοπική κοινωνία και στο πρασίνισμα των πόλεων να σας δώσω μερικά παραδείγματα ε, για το τι κάνει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχουν οι τοπικές ε, αρχές ε, τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρασίνισμα και αυτό είναι προς το καλό όλων και φυσικά και των ανθρώπων που ζουν εκεί. Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί για τη δημιουργία ενός βραβείου που δημιουργήθηκε πριν από 9-10 χρόνια που είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Πόλη. Ε, κάποιος βουλευτής μίλησε για τη Λισαβόνα λέγοντας ότι το 2020 η Λισαβόνα θα είναι η πράσινη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αυτή θα είναι και μια θαυμάσια ευκαιρία να επιμείνουμε στη σημασία για το, το 2020 θα έχουμε τη δεκαετία ε, του βραβείου αυτού τη δέκατη επέτειο από την εγκαθίδρυσή του. Γι' αυτό ε, επιβραβεύει πόλεις ε, που έχουν κάνει προσπάθειες ε, από πολλούς τομείς έτσι ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες. Το ανέφεραν και πολλοί βουλευτές αυτό. Επίσης, θέλουμε να συνεργαστούμε περισσότερο μαζί σας ως θεσμικό όργανο, έτσι ώστε αυτή η εκδήλωση να προβληθεί περισσότερο και να τονίζουμε τη βιοποικιλότητα, τις πράσινες υποδομές, ε, όπως ε, είναι και η βασική εστίαση του ψηφίσματός σας. Θα πρέπει να επιστήσουμε περισσότερο την προσοχή τη σημασία, ε, που, στη σημασία μάλλον που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για το πρασίνισμα του περιβάλλοντος το τονίσατε κι εσείς, η βιωσιμότητα είναι κάτι το εγκάρσιο. Ας πούμε στην ε, ατζέντα, στο θεματολόγιο για τις πόλεις έχουμε ε, πολλές εταιρικέ σχέσεις και συνεργασίες ε, για τη χρήση γης που ανέφερε κάποιος βουλευτής και τη βιοπικιλότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι ένα πρόγραμμα δράσης αυτό τον καιρό στη δημόσια διαβούλευση και θα προτείνουμε και πολλές δράσεις σε όσους παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για να βελτιωθεί η χρήση γης και βιοπικιλότητα. Και φυσικά αυτό θα δώσει λύσεις για τους βασικούς παράγοντες ε, στρες στην πόλη, όπως είναι η ρήπανση, η ρήπανση των υδάτων, της ατμόσφαιρας κτλ. Επίσης και ειδικά εργαλεία χρειάζονται και υπάρχουν ειδικά μέτρα, γιατί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν κάτι που αναφέρατε προηγουμένως, υπάρχουν διάλογοι για τον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει και τις προσφυγές επί παραλήψη, αλλά ε, και φροντίζει να βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις. Το 2016 επίσης άρχισε ένα νέο πρόγραμμα για τις πράσινες υποδομές. Σε 20 πόλεις να συμμετέχουν ε, και συνεχίζεται η συμμετοχή. Επίσης έχουμε ένα κατάλογο 40 ε, πόλεων που ήταν φιναλίστ ή που κέρδισαν το βραβείο της Πράσινης Πόλης για να μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές και οι πόλεις μπορούν να μαθαίνουν, να διδάσκονται η μία από την άλλη και να βελτιώνουν τα πράγματα. Φέτος επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη συμμετοχή, ε, προσοχή μάλλον σε αυτό. Διοργανώσαμε την Πράσινη Εβδομάδα που ήταν αφιερωμένη στο πρασίνισμα των πόλεων. Τεράστια επιτυχία. Και είχαμε και κάποιες συνεδριάσει συνεδριάσεις ή ε, ε, κάποιες συναντήσεις πόλεων που είχαν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να συναντήσουν μια άλλη πόλη και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες. Είναι πολύ σημαντική η τοπική αυτοδιοίκηση. Καλή είναι η επικουρικότητα, αλλά το τοπικό επίπεδο παραμένει. Είναι πολύ σημαντικό και στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βιωσιμότητα ε, εν γέννη επίση ε, είναι κάτι το οποίο ε, διευθύνεται από εκεί και για την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE που στηρίζει τη φύση και την βιοπικιλότητα προτείνεται αύξηση εκεί ε, κατά 25% των πόρων. Με χαρά να συνεχίσουμε τη συνεργασία και τις συζητήσεις μαζί σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. 8 χρόνο διάγραμμα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 14-11 στις 11 η ώρα. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος εδώ στις 6 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας ενώ η συζήτηση και ολομέλεια, και η ψηφοφορία συγγνώμη, στην Ολομέλεια θα πάει το Γενάρη στο Στρασβούργο. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα μας που είναι ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπιόρν Χάνζεν, εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού ΕΧΑ και σας παρακαλώ να έρθετε στο Προεδρείο να καθίσετε κοντά μας. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση. Um, Έχουμε δύο βαριά έγγραφα που μας έχετε μοιράσει, Γενική Έκθεση για το 2017 και ο προγραμματισμός του οργανισμού σας για την περίοδο 2018-2020. Θα σας παρακαλούσα να μας συνοψίσετε τα θέματα αυτά και τα πεπραγμένα και τον προγραμματισμό σε ένα τέταρτάκι, αν ε, γίνεται. Και μετά θα συνεχίσει η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Thank you very, very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση να έρθω εδώ, να έχω διάλογο μαζί σας σχετικά με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών και τις θέσεις του στο ευρύτερο πλήσιο εδώ στην Ευρώπη. Επειδή είναι πρώτη φορά που έρχομαι εδώ, από ό,τι κατάλαβα ο διάλογος αυτός θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ε, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις και κατόπιν να συνοψίσω κάποια από τα θέματα του 2019, αλλά να μιλήσω και για την επόμενη πενταετία ως εισαγωγή στη συζήτηση. Σχεδόν ένα χρόνο βρίσκομαι στη θέση αυτή και σχεδόν πριν ένα χρόνο βρέθηκα εδώ, καθόμουν λίγο πολύ στην ίδια καρέκλα για την ακρόασή μου και είχα διάλογο μαζί σας σχετικά με την θέση μου ως νέου διευθυντή του ΕΧΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών. Και πρέπει να σας πω ότι Πολύ με ενδιαφέρει η επαφή πολιτικής και επιστήμης όσον αφορά τα χημικά και δεν έχω χάσει ούτε ένα γραμμάριο του αρχικού μου ενθουσιασμού ε, και γι' αυτό χαίρομαι που μπορώ να εργάζομαι στην πλευρά των επιστημόνων ενώ παλιότερα εργαζόμουν στην πλευρά των πολιτικών. Δεν έχω χάσει λοιπόν καθόλου τον ενθουσιασμό μου και θα ήθελα να πω ότι Πολύ με βοήθησε ο ίδιος ο οργανισμός, το προσωπικό του, η γραμματεία του, καθώς ε, και ε, τα μέλη του ε, Διευθυντικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Προσφυγών. Όλοι οι συνεργάτες με βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν πολύ υπομονετικοί μαζί μου πέρασα όλα τα κλασικά βήματα. Πρώτα ε, ε, ένιωθα χαμένος, μετά είχα ένα μήνα του μέλητος ε, και τώρα επιτέλους νιώθω ότι κατάλαβα το νόημα και είμαι διατεθειμένος να ηγηθώ του οργανισμού τα επόμενα πέντε χρόνια και να δώσω τις κατευθύνσεις για την επόμενη δεκαετία. Όσον αφορά τις προκλήσεις μας το 2019 και ίσως και λίγο μετά, Καταρχάς, ε, να σας αναφέρω τα ισχυρά μας σημεία, τα πλεονεκτήματά μας ε, και να σας πω πώς πιστεύω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είδα πώς ε, λειτουργούν οι διάφορες επιτροπές, το προσωπικό μας ε, βλέπω ότι ε, ε, έχουν πολλές δεξιότητες οι συνεργάτες μας, καθώς και κατανόηση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί χημικών. Καταλαβαίνουμε καλά τις συνέργειες ανάμεσα στα διάφορα είδη νομοθεσίας και θα γνωρίζετε ότι ο κανονισμός REACH που ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών ε, έχει να κάνει με πολλά άλλα μέρη της νομοθεσίας, ε, μεταξύ των οποίων και νομοθετήματα που δεν ε, εφαρμόζουμε εμείς στη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Έχουμε για παράδειγμα τους πλαστικοποιητές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει νομοθεσία για τα ε, ε, υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Αυτές λοιπόν είναι οι προκλήσεις μας για το 2019 και θα ξεκινήσω λοιπόν ε, από ε, τον ε, κανονισμό REACH καθώς και τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμαση και τη συσκευασία. Και θα σας μιλήσω για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών και για τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε συνοπτικά ότι ε, έχα προχωράει καλά, απομένουν όμως πολλά να γίνουν, μπορεί, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Επίσης, ο κανονισμός REACH είναι αποτελεσματικός, δηλαδή οι μηχανισμοί του πετυχαίνουν τους στόχους τους, αλλά δεν ε, είναι ακόμα ε, απόλυτα αποτελεσματικό. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα, απομένουν πολλά να γίνουν για να πετύχουμε τους στόχους του κανονισμού αυτού. Είχαμε την ε, διάσκεψη ε, κορυφής ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη και έχουμε και στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των χημικών. Οι στόχοι λοιπόν είναι καλοί, αλλά βρισκόμαστε ακόμα πολύ πίσω. Εμείς λοιπόν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς με βάση τις εμπειρίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι μέχρι τώρα ε, για το πρόγραμμά μας για το 2019 και μετά από αυτό. Έχουμε και άλλα νομοθετήματα που εφαρμόζουμε, πέρα από το ΡΙΤΣΕ και την νομοθεσία ενταξινόμηση, την ε, επισήμανση και τη συσκευασία, έχουμε τον κανονισμό για τα βιοκτώνα, που είναι ε, το μικρό αδερφάκι του κανονισμού για τα φυτοφάρμακα. Έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά τις ε, αξιολογήσεις, έχουμε λιγότερες αδειοδοτήσεις και έχουμε εδώ την καινοτομία των βιοκτώνων Έχουμε το, το, την καινοτομία όσον αφορά τα βιοκτώνα σε σχέση με τα φυτοφάρμακα, ότι οι επιχειρήσεις ε, υποβάλλουν αιτήσει για αδειοδότηση, όπως γίνεται και στον κανονισμό REACH, αλλά έχουμε καθυστερήσει, δεν έχουμε αρκετούς πόρους ε, και αυτό λοιπόν αποτελεί μια πρόκληση. Θα πρέπει να επιταχύνουμε. Όσον αφορά τη διαδικασία συνένεσης μετά από ενημέρωση, ε, είναι τεχνικός ο τίτλος, εφαρμόζει όμως ε, την συνθήκη του Ρότερνταμ που μάλλον ε, είναι η πιο αποτελεσματική συνθήκη για τα χημικά που έχουμε. Διασφαλίζει ε, να διαδίδονται οι πληροφορίες σε όλο τον κόσμο για τα επικίνδυνα χημικά και για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Η συνθήκη ήταν πολύ επιτυχής, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι έχουμε περισσότερη δουλειά από ό,τι περιμέναμε. Τα πάμε όμως αρκετά καλά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι η ε, επιτυχία της συνθήκης αυτής είναι ότι βοηθάει τον κόσμο να χειριστεί με ασφάλεια τα πιο επικίνδυνα χημικά. Και για το 2019 και για το μέλλον ε, ο ΕΧΑ έχει αναλάβει νέα καθήκοντα. Είμαι πολύ περήφανος και ευγνώμων για αυτό. Πιστεύουμε όμως ότι και οι δεξιότητές μας για την επίτευξη συνεργειών μεταξύ ε, των καθηκόντων μας, αλλά και για να υπάρχει ε, συνεκτικότητα με τα το κοινοτικό εκτιμένο όσον αφορά τα χημικά αλλά και σε όλο τον κόσμο ε, είναι κάτι που μας ε, ε, κάνει ικανούς να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν την κανονική νομοθετική διαδικασία, έχουμε τον κανονισμό για τους έμονους οργανικούς ρήπους που εφαρμόζει την συνθήκη της Στοκχόλμης, έχουμε τη δημιουργία ενός κέντρου δηλητηρίων όπου εμείς θα είμαστε η σπονδυλική στήλη. Θα επιτρέπουμε θα, θα δίνουμε συμβουλές στα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων για να βοηθήσουν τους πολίτες τι να κάνουν όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, αν κάποιος καταπιεί ένα απορριπαντικό. Επίσης, πρέπει να βοηθάμε τη Γενική Διεύθυνση ε, Απασχόλησης ε, ώστε ε, να έχουμε ε, επίπεδα έκθεσης ε, στην εργασία για τα, χημικά, για τα χημικά και επίσης θα πρέπει να έχουμε μια βάση δεδομένων για τα χημικά και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οδηγίας για τα απόβλητα. Όπως σας είπα, η ανάληψη αυτών των νέων καθηκόντων αποτελεί τιμή, αποτελεί όμως και πρόκληση για το προσωπικό μας. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα, ε, από το 2019, να κοιτάξουμε την επόμενη πενταετία ή δεκαετία, δύο βασικά θέματα θα πρέπει να αναφέρουμε. Ολοκληρώνουμε το στρατηγικό σχέδιο μας ε, που περιγράφει πού θέλουμε να πάμε, ε, τι θέλουμε να κάνουμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Δύο βασικές πρωτοβουλίες βλέπουμε. Η μία είναι να γίνουμε ακόμη καλύτεροι στον εντοπισμό ανησυχητικών χημικών, χημικών που προκαλούν ανησυχίες ε, και να παρέχουμε τις ε, απαραίτητες συμβουλές για το χειρισμό τέτοιων χημικών και η άλλη προτεραιότητα είναι να διασφαλίζουμε την διαβίβαση πληροφοριών ε, σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες στους χρήστες των χημικών και στους καταναλωτές, ώστε να έχουμε ασφαλή χρήση των χημικών. Και η τρίτη προτεραιότητά μας ε, είναι η ε, ολοκλήρωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας πάνω στο ΡΙΤΣΕ και στην, ε, στον κανονισμό CLP, εντάξει νόμιση στην επισήμανση και τη συσκευασία. Ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε οι εργασίες μας πάνω στα χημικά αυτά ε, να περάσει στο γενικό κεκτημένο για τα χημικά, αλλά να χρησιμοποιηθούν και στο διεθνές θεματολόγιο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά. Αυτοί λοιπόν οι τρεις στρατηγικοί στόχοι, αυτές οι τρεις στρατηγικές προτεραιότητες συνδέονται στενά με αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Έκθεση στην, επιτροπή της, στην ε, έκθεσή τη, όπου ε, λέει ότι ε, είναι χρέο μα να διασφαλίσουμε τις συνέργειε αυτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διάθεση επίπεδο. Και τέλο. το τελευταίο μας θέμα είναι το πολιτές πλαίσιο το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή. οργανισμός αυτός ε, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην ε, διασφάλιση υπεραιτέρω συνεργειών ε, και στην εφαρμογή και άλλων νομοθετημάτων. Εάν λοιπόν αυτό αποτελέσει απέτηση από εσά και από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα περιμένουμε και σταθερή χρηματοδότηση εντός του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε τη σύνδεση των δικών μας εργασιών ε, με ε, άλλα νομοθετήματα τα οποία δεν εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή, για τα οποία όμως έχουμε γνώσεις ε, και δεξιότητες. Με αυτά τα λόγια λοιπόν θα ήθελα να κλείσω την εισαγωγή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και προσβλέπω στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στο άτομο επαφής τη Επιτροπής μας, ε, τον κύριο Πιερά. Ε, το άτομο επαφής με την ECHA. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλώς ορίσατε κύριε Δευθυντά και ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας. Την 1η Ιανουαρίου του 2018 γίνατε διευθυντής. Ε, έχετε λοιπόν τη θέση αυτή εδώ και περίπου 10 μήνες. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα, αλλά αρκετό για να πει κανείς ότι έχετε αποκτήσει μια εικόνα των δραστηριοτήτων τη ECHA και ε, μια εικόνα του τι πρέπει να γίνει. από ό,τι κατάλαβα θέλετε να εστιαστείτε στις ε, κυρίες στρατηγικές, ε, ειδικότερα για παράδειγμα στο ζήτημα της ε, ανταλλαγής πληροφοριών περί χημικών προϊόντων. Εμείς θέλουμε η ΕΚΑ να είναι και επιστημονικό κέντρο το οποίο θα μπορεί να ασχοληθεί με κάποια ζητήματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης ε, των χημικών προϊόντων. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπατε. Το συζητήσαμε και νωρίτερα σήμερα το πρωί. Εμένα θα με ενδιαφέρε να ακούσω περισσότερα όσον αφορά τα συμπεράσματα για τον κανονισμό REACH και για τις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού. Ειδικότερα όσον αφορά τη δημιουργία νέων, μιας νέας βάσης δεδομένων. Θα με ενδιαφέρει επίσης να ακούσω και πληροφορίες για τους ε, δυνατούς ε, τρόπους δημιουργίας κέντρων, αποθήκευσης ε, δηλητριωδών και βιοκτώνων προϊόντων. Το 2018 είναι σημαντική χρονιά είναι το έτος ε, στόχος για τα δεδομένα καταγραφής όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές για τις εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείε. Εισαγωγές εξαγωγές άνω των χίλιων τόνων χρειάστηκε να καταγραφούν όσον αφορά τα χημικά στα οποία αναφερόμαστε. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μάθω τι ουσίες έχουν εξαχθεί προς ποιες χώρες και σε τι ποσότητες. Η διαφάνεια πιστεύω είναι κλειδί. Επίσης θα ήθελα να μάθω περισσότερα όσον αφορά την ε, καταγραφή και έγκριση εισαγόμενων χημικών στην Ευρώπη. Η ποιότητα επίσης των πληροφοριών καταγραφής είναι σημαντική. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, το 1 τρίτο των χημικών που εγκρίνονται για εισαγωγές ε, στην Ευρώπη, για προσαγωγές στην Ευρώπη, είναι αμφιβόλου ασφαλείας. Κάποιοι μάλιστα αναφέρονται σε ανεξέλεγκτες εισρωές χημικών προϊόντων στην Ευρώπη. Η ΕΚΑ πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το μέτωπο και να συνεργαστεί με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ως πολιτικός επίσης και, αλλά και ως ε, γιατρός θέλω να τονίσω ότι δεν μπορούμε να υποτιμάμε ε, και να υπονομεύουμε την ανθρώπινη υγεία. Το βάρος τη αποδείξη το φέρνουν οι επιχειρήσεις. Αυτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα χημικά που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή. Σύμφωνα ωστόσο με το Γερμανικό Οργανισμό Χημικής Ασφάλειας, το 1 τρίτο των χημικών που καταγράφονται ε, στο πλαίσιο του REACH δεν συνοδεύονται από αξιόπιστες εκθέσεις ασφαλείας. Αυτό ε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στον πολιτικό διάλογο και στις δραστηριότητες ε, της ΕΚΑ. Ναι, εντάξει, ξέρω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες εντός της ΕΚΑ αλλά και από τον κόσμο γενικότερα. Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στρατηγική πιο διαφανή αν το 1 τρίτο των χημικών δεν συνοδεύεται από μελέτες, δεν τεκμηριώνεται από μελέτες ασφαλείας. Η ανυπαρξία μελετών δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή τα προϊόντα αυτό. Αυτό δεν ε, συνάδει με τον κανονισμό REACH. Πρώτα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε ε, στην ακριβή καταγραφή. Εφόσον η καταγραφή δεν έχει γίνει με τον σωστό τρόπο, η υπόλοιπη διαδικασία δεν θα πρέπει να μπορεί να ολοκληρωθεί με θετική απόφαση κυκλοφορίας ε, στην αγορά. Η διαφάνεια λοιπόν όλων των δεδομένων για παράδειγμα για επιχειρήσεις που δεν έχουν παρασχεί πλήρη τεκμηρίωση είναι κάτι απολύτως αιτιολογημένο. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να γίνεται και δημόσια αυτό. Ε, να δημοσιοποιούνται δηλαδή αυτές οι πληροφορίες. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το περιεχόμενο ορισμένε φορές, αλλά είναι ύψης της σημασίας ε, η αξιοπιστία της ΕΚΑ. Η ΕΚΑ θα πρέπει να εργάζεται προς όφελος ε, και των ανθρώπων και των επιχειρήσεων ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, καλώς ορίσατε κύριε Πρόεδρε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ο Γερμανικός Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και το BFR που είναι πολύ γνωστό από την περίπτωση Glyphosat σας έχουν επιτεθεί σφοδρά. 100.000 ε, μόρια χημικές ουσίες κυκλοφορούσαν στην Ένωση. Συστήθηκε ο Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ΕΧΑ. Από το 2007 έπρεπε να κάνετε μια αξιολόγηση. Πού βρισκόμαστε. Από το 2015 και μετά οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση με φάκελο για την καταχώρηση. Άκουσα ότι ε, από το 8 ε, μέχρι το 17 είχατε 1952 φακέλους. Όπως είπε και ο συνάδελφος, μαθαίνουμε ότι το 1 τρίτο ε, δεν συμμορφώνεται ή δεν έχει ελεγχθεί. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό. κάτι άλλο που μας ανησυχεί. Ε, και αφορά την ε, επιτροπή μας PEST ε, και σας αναφορά και σας. Εγώ κατασκευάζω μια χημική ή παρασκευάζω ουσία και σας στέλνω ένα φάκελο. Τι κοιτάτε, όλες τις μελέτες. Εγκρίνετε την ενέργεια ουσία για να κυκλοφορήσει στην αγορά και εκ των υστέρων πάτε να διασταυρώσετε επί της ουσίας αν ο φάκελός μου είναι πλήρης και ποια είναι η τοξικότητα των προϊόντων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για σας όμως, διότι με την καταχώρηση ε, και την καταγραφή επιτρέπεται στον κατασκευαστή να πουλάει τα προϊόντα του και να τα διαθέτει στην αγορά και μετά διαπιστώνουμε ότι «Α, μα είναι άκρος τοξική αυτή η ουσία». Και στον κανονισμό λέτε ότι υπάρχει 5% υποχρέωση ε, ανάλυσης των δειγμάτων. Γιατί να το αυξηθεί αυτό, γιατί 5%, το 100% να ελέγχεται. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, όπως είπε ο συνάδελφος, είπατε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Ωραία. Πόσα και πόσους εμπειρογνώμονες. Γιατί θα πρέπει να μιλάμε μετά με συγκεκριμένο τρόπο κάποια στιγμή. Για τα βιοκτώνα τώρα. Έχω μάθει, έχει φτάσει στα αυτιά μου, και θέλω να μου πείτε τη θέση σας, ότι όταν υπάρχουν ομάδες αξιολόγησης για τα βιοκτώνα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προσκαλείται και τη βιομηχανία. Γιατί καλείται τη βιομηχανία. Γίνεται ολόκληρη αντιπαράθεση για τη σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Όταν έχετε τα βιοκτώνα να αξιολογήσετε, να έρχονται οι από τα κράτη-μέλη, τι δουλειά έχουν οι βιομηχανίες εκεί πέρα μέσα στις ομάδες εργασίας. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω και συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως ήταν συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον ΕΧΑ. Δεν είναι αυτό. Και αν, χρειάζεται, αν χωράει βελτίωση, τώρα πρέπει να γίνει. Να δείτε στους βουλευτές, κοιτάξτε ποιες είναι οι δυσλειτουργίες, τα προβλήματα, τι μας χρειάζεται για να βελτιωθούμε. Η έκθεση BFR είναι πολύ σκληρή ε, για αυτά που κάνατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγχαουτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Χάνσεν για την εισαγωγή του. Από τις ερωτήσεις βλέπετε ήδη ότι μας εκπλήσει κάπως ε, η εισαγωγή σας και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ έχω εκπλαγεί. Γιατί ξέρετε ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορες πληροφορίες και τώρα θα μας πείτε ότι αυτά ήταν γνωστά και δεν ήταν καμιά είδηση και δεν βελτιώνει την κατάσταση ή δεν την επιδεινώνει. Εγώ θα σας πω ότι αυτό παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχει να κάνει με την ίδια την ίδρυση και λειτουργία του REACH. Άρχισε από το 2007 και μέχρι το 2010 ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι και είναι αρμόδιος οργανισμός ΕΧΑ για να τα ελέγξει όλα αυτά. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα και πλέον, ε, αν έρθουμε στο συμπέρασμα ότι το 1 τρίτο των φακέλων για τις χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ε, τότε έχει αποτύχει απλούστατα ο οργανισμός σας. Ακόμα και μας λέτε ότι μπορούμε να ελέγχουμε μόνο 5% ή αυτό επιβάλλει ο νόμος. Πόσοι είναι οι φάκελοι, πάνω από 40.000. Και το 5% πόσο είναι. Πόσες άδειες έχετε ανακαλέσει, 4, 5. Αυτό είναι πολύ λιγότερο από το αν κάνατε πραγματικό έλεγχο του 5%. Και η οδηγία REACH είναι ξεκάθαρη. Όταν δεν δίνει στοιχεία, δεν σου δίνεται η άδεια να κυκλοφορεί στην αγορά. No data, no market. Και αν το 1 τρίτο των χημικών ουσιών δεν έχουν πλήρη φάκελο και δεν υπάρχουν δεδομένα, τότε τι δουλειά έχουν να κυκλοφορούν στην αγορά. Και παρόλα αυτά κυκλοφορούν όλε οι ουσίες. Ε, τι έχει κάνει ο οργανισμός ΕΧΑ. Εκτό από το να λέει το φάκελο δεν είναι πλήρη και να το επιστρέφεται στι εθνικέ αρχέ. Τώρα σε αυτό το παιχνιδάκι θα μπούμε στην κολοκυθιά που θα παίζετε με τις εθνικές αρχές εσείς και ευρωπαϊκές, έτσι θα εμπιστευόμαστε τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είναι ευθύνη του οργανισμού σας. Όταν κάποιος δεν δίνει στοιχεία, ε, δεν παίρνει άδεια να κυκλοφορεί στο προϊόν στην αγορά. Έχει έρθει η ώρα να υψώσετε το ανάστημά σας και τη φωνή σας και ο οργανισμός και εσείς και να δείξετε πόσο σας καίει αυτό το θέμα και πόσο επίγον είναι και σας ανησυχεί. Και δεν αρκεί να πούμε ότι δεν είναι ασφαλή τα χημικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το ξέρουμε και είναι χημικά που κυκλοφορούν ευρύτατα, το 95% του όγκου που κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Και για το 1 τρίτο δεν ξέρουμε για την οικοτοξικότητά τους, αν είναι πλήρης η φάκελη, όχι. Ίσα ίσα ξέρουμε ότι δεν είναι πλήρης, άρα δεν έχουν γίνει κάποιες μελέτες. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αρχίσετε να τα λέτε όλα αυτά ξεκάθαρα, για ποιες δράσεις έχετε αναλάβει, για ποιους φακέλους και για ποιο λόγο κυκλοφορούν ακόμα τα προϊόντα. Και τι να τα κάνω τα μνημόνια που βγάλατε το καλοκαίρι, όταν πάλι μιλάτε για την ποιότητα των δεδομένων. Αυτά είναι λόγια που ακούμε χρόνια τώρα από την ΕΧΑ. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα. Είναι ότι δεν έχουν δεδομένα, δεν τα έχουν δώσει οι άνθρωποι. Και είναι το REACH, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εσείς πρέπει να κάνετε κάτι, εσείς είστε υπεύθυνοι. Και όταν λέτε χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό, πόσου θέλετε παραπάνω. Γιατί δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από αυτό. Η ε, ασφάλεια των πολιτών που θα πρέπει να ξέρουν 100%, εντάξει, 100% υπερβάλλω, δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Αλλά να είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι πλήρη η φάκελη και οι αιτήσει, γιατί αυτό απαιτεί ο νόμο και δεν είναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο οργανισμό ΕΧΑ τώρα μας λέει χρόνια ολόκληρα ότι θέλει να το βελτιώσει, αλλά το μόνο που βλέπουμε είναι μνημόνια που κάνετε με τη χημική βιομηχανία. Και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και μας λένε, για να είμαι ειλικρινής, σκοτίστηκα. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αυτοί θα πρέπει να δώσουν τα δεδομένα και να είναι πλήρη η φάκελη. Είναι δική τους υποχρέωση και δική σας υποχρέωση είναι να τηρούν ε, τον νόμο, αλλιώς τους αφαιρείτε την άδεια. Δυστυχώς όμως κυκλοφορούν ακόμα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας και πρέπει να το λύσετε και γρήγορα. Και μην ακούμε άλλο ένα χρόνο λόγια και μνημόνια συνεννόησης με την χημική βιομηχανία. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μάρτιν εάν έχει κάποιες παρατηρήσεις. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο. Η δόκτωρ Μάρτιν είναι η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διευθυντικό Συμβούλιο του ΕΧΑ. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω που με ορίσατε εκπρόσωπό σας στο Διευθυντικό Συμβούλιο του ΕΧΑ. Αυτό το πρώτο έτος ήταν έτος εορτασμών ε, αλλά και προκλήσεων. Το 2017 ξεκινήσαμε και πρέπει να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Ε, εντός των 28 κρατών ε, μελών ε, το REACH ήταν πολύ σημαντικό βήμα και έχει αποτελέσει και υπόδειχνα για άλλες χώρες όπως είναι η Κίνα, η Κορέα, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία. Το 2017 ήταν και το έτος προθεσμίας ε, για την καταχώρηση ε, ουσιών και ως ε, Ευρωπαία που έμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο εντυπωσιάστηκα από τις εργασίες αυτές. Ήταν έτος αλλαγών και έχουμε και νέο εκτελεστικό διευθυντή αλλά απομένουν πολλές προκλήσεις. 22.000 ουσίες έχουν ε, καταχωριστεί, απαιτούνται όμως προσπάθειες για να ε, σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο. Τέλος, ε, ο ΕΧΑ έχει αναλάβει και νέα καθήκοντα. Θα πρέπει να δημιουργήσει νέα βάση δεδομένων για την παρουσία επικίνδυνων ουσιών και ως ε, πολίτης αλλά και ως ερευνήτρια επικροτώ αυτήν τη νέα πρωτοβουλία. Πολλά μπορούμε να μάθουμε από ε, περαιτέρω ε, έρευνα των τεχνολογιών ανακύκλωσης αναλύοντας τη σύνθεση των αποβλήτων. Πιστεύω ότι ο ΕΧΑ έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα. Χρειαζόμαστε όμως ε, την υποστήριξη των θεσμικών οργάνων ε, και την ε, σχετική χρηματοδότηση. Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες θα προσπαθήσω να απαντήσω στο βαθμό που είναι δυνατόν και θα μπορέσω να σας κατευθύνω και προς άλλες πηγές πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα παρακαλούσα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο εάν έχει παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάντσεν αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία. Όσον αφορά τα πρόσθετα καθήκοντα και τους πόρους, ε, συνεργαζόμαστε στενά με την ΕΚΑ, ώστε να θεωρούμε ότι θα παραμείνει επιχειρησιακή ακόμη και με τα νέα καθήκοντα που τις ανατίθενται. Αυτό γίνεται όχι μόνο με τις ε, Λειτουργικέ Υπηρεσίε Κομισιόν αλλά και με την ε, δημοσιονομική υπηρεσία της Κομισιόν για τις άλλε πτυχέ ε, για την καταγραφή, για τη συμμόρφωση. Όλα αυτά έχουν ήδη εντοπιστεί μέσω της ε, αναθεώρησης που υιοθετήσαμε και υποβάλαμε στο Κοινοβουλίο την Άνοιξη φέτο. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τι δράσει. Όχι μόνο όσον αφορά την καταγραφή, την εγγραφή, αλλά και όλα τα θέματα σε συνεργασία με την ΕΚΑ, τα κράτη-μέλη και του εμπειρογνώμονε. Είναι φυσικά ανησυχητικά κάποια στοιχεία. Ε, κάτι που υπογραμμίζει περισσότερο ακόμα την ανάγκη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο θέμα αυτό και αν χρειαστεί να πάμε και πιο πέρα από τα καθήκοντα που έχουμε ε, προβλέψει στο ΡΙΤΣ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρο. Ακούσαμε κάποιε ενδιαφέρουσε ερωτήσει και παρατηρήσει. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Χάντσεν, εκτελεστικό διευθύντη τη ε, ε, ΕΚΧΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, ώστε να απαντήσει τι ερωτήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω πράγματι να δώσω κάποιες απαντήσεις και σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολλές σας ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη αν οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ε, δεν ε, περιέγραψαν λεπτομερώς όλα τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επέλεξα από έναν πολύ μεγάλο κατάλογο να αναφερθώ στη δεκαετή έκθεση της Κομισιόν που περιλαμβάνει επίσης ένα τεράστιο κατάλογο πραγμάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οπότε θέλω να σας δηλώσω εδώ ότι δεσμεύομαι να τα αντιμετωπίσω όλα. Όσον αφορά το ζήτημα τη συμμόρφωση, να κάνω κάποιε αρχέ παρατηρήσει και μετά θα προσπαθήσω να απαντήσω με κάποια λογική σειρά. Και για το ζήτημα τη συμμόρφωση θα αναφερθώ πιο λεπτομερό στο τέλο. Αλλά πρέπει να σας πω ξεκινώντας ότι ναι, η ΕΚΑ ε, θα επιταχύνει ε, τι εργασίε τη. Το θεωρώ ότι είναι δικό μου καθήκον να επιταχύνουμε διαρκώ τι εργασίε μα, όπω έκανε και ο προκατοχό μου στον οργανισμό. Είναι καθήκον μου και δουλειά μου. Και σα διαβεβαιώ ότι ούτω θα πράξουμε. Ανησυχία, ναι, ανησυχούμε με, από τα αποτελέσματα της μελέτης BFR. Ε, επιβεβαιώνουν μελέτες ε, και πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και εμείς εσωτερικά. Και πράγματι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το να μην κρυβόμαστε Φυσικά και όχι. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα βρίσκομαι εδώ και γι' αυτό απαντάω όσο μπορώ πιο ευθέω και αν δεν απαντήσω ευθέω παρακαλώ να μου γράψετε για να δεν έχω κανένα σκοπό να κρυφτώ. Να ξεκινήσω με το υπόβαθρο και θα πάω στην καταγραφή αργότερα. Πάμε στο υπόβαθρο. Θα μιλήσω για τις βάσεις δεδομένων, για την καταγραφή, για την εγγραφή αν θέλετε των προϊόντων, για τις βιοεπιστήμες και μετά θα πάω στο ζήτημα του Μνημονίου Συνεννόησης με τη βιομηχανία και ο δικό τους ρόλο στο δικό μας έργο που επιτελούμε για θέματα συμμόρφωσης και μετά μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση αν ε, οι απαντήσεις μου σας αρκούν. Ε, δεν σας αρκούν, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς και το λέω εμείς, ε, όχι εσείς θεσμικά, εμείς στην ΕΚΑ, στην Κομισιόν, όταν ε, σχεδιάζουμε κρατώντας, ε, όταν σχεδιάσαμε το REACH στην Κομισιόν, είχαμε να κάνουμε κάποιες θεμελιώδεις επιλογές όσον αφορά το μοντέλο το οποίο θέλαμε να υλοποιήσουμε. Τα μοντέλα τα οποία είχαμε ήταν το υπάρχον σύστημα, τα υπάρχοντα χημικά που κατά 99% ήταν αυτά που κυκλοφορούσαν στην αγορά και, το, και αυτά που κυκλοφορούσαν στην αγορά κατά 99% μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως είχαν, χωρίς κανένα αριθμιστικό πλαίσιο όπως ήθελε η βιομηχανία. Το άλλο άκρο ήταν ένα σύστημα εξουσιοδότησης όπου οι βιομηχανίες έπρεπε να υποβάλουν φακέλους που θα έλεγχε μια αρχή και ο έλεγχος θα οδηγούσε στην ε, πρόσβαση στην αγορά. Ο έλεγχο θα αφορούσε το κατά πόσο συμμορφώνονται με τι απαιτήσει οι φάκελοι και μετά από τον έλεγχο συμμόρφωση θα ακολουθούσε η άδεια κυκλοφορία στην αγορά. Τα νούμερα που θα σα δείξω όσον αφορά την καταγραφή πάνω από 20.000 ουσίε. Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη λύση, το σύστημα εξουσιοδότηση όπου θα ελέγχαμε εκ των προτέρων τη συμμόρφωση για 20.000 ουσίε πριν του δώσουμε άδεια κυκλοφορία στην αγορά, θα απαιτούσε είτε πάρα πάρα πολλά έτη, πολλά περισσότερα χρόνια από ότι αυτή τη στιγμή, για να τα διεκπαιρεώσουμε όλα, για τι βιοεπιστήμε. για παράδειγμα, καταφέραμε 30 ουσίες, για τα βιοκτώνα, συγγνώμη, καταφέρουμε 30 ουσίες ετησίως και έχουμε 20.000 ουσίες στο REACH. Η απόφαση λοιπόν τότε που έλαβαν υπεύθυνοι χάραξη πολιτική ήταν ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ένα σύστημα εξουσιοδότηση. Οπότε αποφασίσαμε μια υβριδική λύση. Τι να κάνουμε, δηλαδή η βιομηχανία θα πρέπει να υποβάλει τους φακέλους οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρεις και εκ των υστέρων ο οργανισμό ε, επαληθεύει τη συμμόρφωση. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εκ των υστέρων ελέγχουμε τη συμμόρφωση. Και εκεί δεν σας το κρύβω, σας το επιβεβαιώνω και συμφωνώ, ναι ε, ανησυχώ. Το σύστημα όμως έχει δημιουργηθεί ώστε να παραμένουν οι επιχειρήσεις στην αγορά. Δεν είναι στην αγορά δηλαδή παράνομα. Το σύστημα έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρης όλοι αυτοί οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί αλλά ένα μεγάλο κομμάτι τους δεν συμμορφώνεται. Θα μπω στις λεπτομέρειες αυτού του προβλήματος λίγο αργότερα. Να σας δώσω κάποια νούμερα. Εάν Έχουμε πάνω από 20.000 ουσίες, όπως είπαμε, στην ευρωπαϊκή αγορά που έχουν εισαχθεί σταδιακά στο σύστημα REACH. για όλες τις ουσίες αυτές έχουν υποβληθεί πλήρης φάκελοι καταγραφής. Τι είναι οι φάκελοι αυτοί. Είναι τα τεκμήρια που δείχνουν πώς ρυθμίζουν τα χημικά οι ίδιες οι βιομηχανίες. Και τώρα εναπόκειται σε εμά να ρίξουμε μια ματιά σε αυτούς τους φακέλους καταγραφής και να τους πούμε κατά πόσο είναι σωστή η ρύθμιση ή αν σε κάποια πράγματα πρέπει να παρέμβουμε και όπως είπε και ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο, έχουν περάσει οι προθεσμίες, όλοι οι φάκελοι τώρα είναι στο σύστημα, ρυθμίζονται, βρίσκονται υπό ρυθμισή, όλες οι ουσίες αυτή τη στιγμή έχουμε καλύτερη προστασία στην εσωτερική αγορά από ό,τι είχαμε στο παρελθόν, που δεν υπήρχε καθόλου σύστημα. Ωστόσο, εξακολουθούμε να μην έχουμε επιτύχει τον απότερο στόχο μας. Ε, πάμε να δούμε τις βάσεις δεδομένων. Μία από τις αρμοδιότητές μας που ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς ε, και είμαι ευγνώμων όχι μόνο για το προσωπικό της ΕΚΑ ε, και το Διοικητικό Συμβούλιο που το ενέκρινε, αλλά και, για προ... και προς τον προκάτοχό μου, που ανέπτυξε πληροφοριακά τον οργανισμό μας. Είμαστε λοιπόν ένας οργανισμός ε, που χρησιμοποιεί την πληροφορική σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε δυνατότητα διεκπαιρέωση μεγάλου βαθμού δεδομένων και κοινοποίηση των δεδομένων αυτών στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, ενημέρωση πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ αποτελεσματικά, με ελάχιστη ε, ανθρώπινη παρέμβαση. Χάρη σε αυτές τις δυνατότητες μας ανατέθηκε ε, η δημιουργία διαφόρων βασών δεδομένων, όπως ανέφερα η βάση δεδομένων του κέντρου ε, δηλητηριάσεων. Υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες τη εβδομάδα να μπορούν να διαθέτουν hotlines για να βοηθούν ε, του ε, πολίτε όταν έχουν πρόβλημα με κάποια χημικά ή με κάποια δηλητηρία στα κατοίκων. Επίση, εξετάζουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αναπτύξουμε μια βάση δεδομένων για την οδηγία, για το πλαίσιο ε, απορριμμάτων. Εκεί ανοιχνεύονται χημικά, υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού ροών ανακύκλωση. Υπάρχει και η δυνατότητα για όσους παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα να ξέρουν ποιο κομμάτι του προϊόντος τους μπορούν να αναπτύξουν ε, Χωρί ε, ανησυχητικά χημικά. Μιλάμε για μια βάση δεδομένων δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει την καινοτομία αλλά και όσου ε, πραγματοποιούν την ανακύκλωση. Αυτό είναι ένα από του τομεί, ή μάλλον ο τομέα όπου αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Κομισιόν για να διασφαλίσουμε επαρκείς πόρου. Δυστυχώ μια τροπολογία τη επιτροπή σα που παρουσιάστηκε και στην Ολομέλεια που θα μας πάρει είχε περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους, γι' αυτό ε, τα καθήκοντα δεν εγκρίθηκε στην Ολομέλεια. Αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε λοιπόν. Προσπαθούμε να βρούμε του πόρου που χρειάζονται για να δημιουργήσουμε αυτή τη βάση δεδομένων ε, για την ανακύκλωση ε, που ήταν ιδέα του δικού σα κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. ουσιαστικά ε, δημιουργώντα αυτές τις διαφορέ βάσεις δεδομένων, τι κάνουμε, δημιουργούμε συνέργειες, χρησιμοποιούμε δηλαδή ε, κάποιες υποδομές που υπήρχαν ήδη, σημαντικές ποσότητες δεδομένων, γνώσεων, ε, υλικού, υπολογιστών ε, που έχουμε ήδη. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα φθηνότερα από ό,τι αν γίνονταν κάπου αλλού. Πάμε να δούμε τα θέματα διαφάνειας και της βιοεπιστήμης. Ε, και συγγνώμη και τα βιοκτώνα ταυτόχρονα. Χάρη στην ε, πληροφορική όπως τη χρησιμοποιούμε, καταφέρνουμε με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, με δύο ανθρώπους ουσιαστικά χρησιμοποιούμε ε, σε πλήρη απασχόληση για να δημοσιοποιούμε χιλιάδες και χιλιάδες φακέλους στο διαδίκτυο κάθε χρόνο χάρη στην υποδομή πληροφορικής που έχουμε. Να εξοδέψαμε κάποια ευρώ παραπάνω, αλλά έχουμε μόνο δύο άτομα και δημοσιεύουμε, θα μπορούσα να σας πω το 99% των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Η βιομηχανία απαιτείται να υποβάλει αιτήματα εμπιστευτικότητας για τις πληροφορίες και να καταβάλει κάποιο ε, τίμημα γι' αυτό. Ε, και εμείς εξετάζουμε κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι με το αίτημα εμπιστευτικότητας και ε, αν όχι δημοσιεύουμε τις πληροφορίες. Μόνο ένα-δυο φάκελοι έχουν ε, εγκεκριμένα τέτοια αιτήματα εμπιστευτικότητα. Μάλλον ελάχιστα ήταν τα αιτήματα εμπιστευτικότητα από τη βιομηχανία επιλογή. Περισσότερε πληροφορίε δημοσιοποιούνται στο Ιντερνετ. Κατά συνέπεια, αν υπάρχει κάποιο φάκελο με μη συμμορφούμενα δεδομένα, αυτό μπορεί να το δει ο καθένα. Αρκεί να πάει στην ιστοσελίδα μα, να ψάξει να βρει το όνομα τη εταιρεία και τα σχετικά δεδομένα. Εμεί οι ίδιοι δεν πάμε να πούμε ότι δεν είναι συμμορφούμενο ε, ένα φάκελο ή κάποιο άλλο, δεν είναι ρόλο μα αυτό, αλλά παρέχουμε όλε τι πληροφορίε ώστε να μπορεί να πάει οποιοδήποτε θέλει να βρει τα στοιχεία μαζί με τα ονόματα των εταιριών. Για τα βιοκτώνα, τα οποία σχετίζονται με τη διαφάνεια και με παρουσία τη βιομηχανία, ναι, είχαμε τη βιομηχανία. Παρουσίας, ε, τη βιομηχανία παρούσα, αλλά είχαμε παρόντες και πολλούς άλλους ενδιαφερομένους. Είχαμε ε, προσκαλέσει τις πράσινες ΜΚΟ, καταναλωτέ, καταναλωτές, εργαζομένου με ένα σωρό άλλου ενδιαφερομένους. Και εδώ κατά βάση ακολουθούμε τις κατευθυντήριε οδηγίε της Κομισιόν για τι ομάδε. εμπειρογνωμόνων. Προσπαθούμε να έχουμε μια εξισορροπημένη εκπροσώπηση απόψεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση. Ωστόσο, ε, περιοριζόμαστε σε αυστηρά επιστημονικές συζητήσεις. Αν υπάρχει λοιπόν κάποιο πολιτικό μήνυμα ε, δεν το ακούμε. Ε, διακόπτουμε μάλιστα και τους ομιλητές στο μέσο της ομιλίας τους. Μα ενδιαφέρει δηλαδή μόνο η επιστημονική και τεχνική πτυχή. Γιατί έχουμε την παρουσία τη βιομηχανία πολύ συχνά στα βιοκτώνα. Αυτό αποτελεί αίτημα των βιομηχανιών. Ε, μερικές φορές τα αιτήματα των βιομηχανιών δεν είναι απόλυτα σαφή, οπότε χρειαζόμαστε την παρουσία μας για να μας εξηγήσουν τι έχουν ζητήσει, τι κάνουν ε, σε ένα σημείο, σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να μην περνάμε πάλι από γραπτή διαδικασία για να πάρουμε παραπάνω πληροφορίε. Αυτό όμω δεν γίνεται και κλεισμένο των θυρών με τη βιομηχανία, γίνεται ανοιχτά, δημοσίω με όλου του ενδιαφερομένου και φυσικά και με του εμπειρογνώμονε των κρατών μελών. Πάμε τώρα στην ε, μελέτη VFR και στη συμμόρφωση. Να σας δώσω κάποια νούμερα. Διότι έχει γίνει δουλειά. Ε, δεν το λέω αμυντικά ε, ό,τι λέω. Κάνουμε ελέγχους συμμόρφωσης και έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Αλλά αυτές οι προσπάθειες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δεν είναι επαρκείς. Δεν, δεν αρκούν. Αλλά έχουμε εξετάσει 700 ουσίες μέχρι στιγμής. Και για αυτές τις 700 ουσίες έχουμε εξετάσει όλα τα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν στον προσδιορισμό της ουσίας ως ουσίας πολύ Έχουμε εξετάσει λοιπόν 700. Από αυτές τις 700 τα 2 τρίτα καταλήγουν ε, να πούμε, καταλήγουμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε. Δηλαδή, τα στοιχεία που έχουν δώσει οι βιομηχανίε, κατά την άποψή μα, δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό REACH. Συνεπώ, απαιτούμε να γίνουν δοκιμέ ε, συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH για τα δύο τρίτα των περιπτώσεων. Αλλά στην προσέγγιση μας δεν πάμε να επιλέγουμε τυχαία κάποιες ε, ουσίε, επιλέγουμε τις ουσίε εκείνε που είναι πιο πιθανό να μην συμμορφώνονται με τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή ε, τα εργαλεία IT που έχουμε, χάρη ε, στην υπηρεσία μας IT, μπορούμε εύκολα και με μεγάλη επιτυχία να βρούμε τις ουσίες που είναι πιθανότερο να μην συμμορφώνονται και επίση ε, εκείνες που ε, χρησιμοποιούνται σε υψηλότερη ποσότητα, σε μεγαλύτερη έκθεση, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση. Όπω είπα λοιπόν όμως ε, και αυτές τα δύο τρίτα απαιτούν περισσότερε προφορίες. Ακολουθούμε τον κανονισμό REACH, αλλά αυτό δεν είναι σύστημα εξουσιοδότηση όπω εξηγήθηκε εδώ. Δεν μπορούμε εμεί να φτιάξουμε κάποιο σύστημα εξουσιοδοτήσεων, διότι θα απαιτούσε υπερβολικά πολλή δουλειά. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καλύψουμε τα κενά, την καθυστέρηση που έχουμε σε θέματα συμμόρφωση. Αυτά όσον αφορά τα νούμερα. Τι κάνουμε εμείς. Ναι και εγώ ανησυχώ πράγματι και το προσωπικό μου ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2019, κάτι που θα συζητηθεί και που θα πρέπει να υιοθετηθεί στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου το Δεκέμβριο και σαφώς το ζήτημα της συμμόρφωσης έχει υψηλή προτεραιότητα. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν προηγουμένως ε, αναφέρεται αυτό ήδη στην αναθεώρηση της Κομισιόν. Το ετοιμάζουμε λοιπόν εν ώψη του 2019 ως θέμα ύψης της προτεραιότητας. Τι σημαίνει αυτό, ότι χρειάζεται να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή να του δώσουμε προτεραιότητα, να δώσουμε περισσότερους πόρους και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά ήδη εδώ πολλά χρόνια και σα το λέω και από προσωπική μου εμπειρία, του τελευταίους 10 μήνε, εξετάζουμε το πώ η διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, στον οργανισμό μα ε, μπορεί να γίνει ταχύτερη, ε, διατηρώντα ταυτόχρονα την νομική και επιστημονική τον νομικό και επιστημονικό έλεγχο σε ικανοποιητικό επίπεδο, σε επαρκέ επίπεδο. Δηλαδή να κάνουμε τα ίδια με περισσότερου πόρου, αλλά να βάλουμε και περισσότερου πόρου για να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Για να σα δώσω μερικού αριθμού τώρα, όπω ζητήσατε με ένα μέλο του προσωπικού σε πλήρη απασχόληση μπορούμε να κάνουμε πέντε ελέγχου συμμόρφωση. Μπορούμε να εξετάζουμε δηλαδή πέντε φακέλου με κάθε ένα άτομο ε, σε διάστημα ενό έτου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε τελική ανάλυση, εγώ εκπροσωπώ τον οργανισμό αυτό και βρίσκομαι εδώ για να εξυπηρετήσουμε εσά. Μπορούμε να κάνουμε του υπολογισμού μαζί. Αν θέλετε 100% όλων των χημικών ε, που χρησιμοποιούνται σε υψηλές ποσότητες μπορούμε να καθίσουμε κάτω και να σας πω πόσο καιρό θα χρειαστεί με τους σημερινούς πόρους. Μπορώ να σας πω, ελπίζω να γινόμαστε όλο και πιο αποτελεσματικοί ε, και έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι που δουλεύουν για μένα αποκτούν όλο και περισσότερες γνώσεις, όλο και μεγαλύτερη εμπειρία, οπότε μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά Βάσει αυτό μπορώ να σα πω εγώ πότε μπορούμε να τελειώσουμε, μπορείτε να μου πείτε εσείς πότε θέλετε να τελειώσουμε και θα, τότε θα σα πω εγώ τι πορεία χρειάζονται. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαι περισσότερα ε, από τη μία σελίδα που έχω μπροστά μου. Χρειάζομαι ένα εξελόφυλλο στο κομπιούτερ, αλλά ευχαριστώ να σα δώσετε τι πληροφορίες αν μου το ζητήσετε. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω ξανά είναι προτεραιότητα για μας. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε εσά του πολίτε και φυσικά το θέμα αυτό ε, δημιουργεί κάποιες ανησυχίες, οπότε θεωρούμε ότι χρειάζεται προτεραιότητα ε, για το 2019. Το μνημόνιο συνενώσεις που έχουμε με το ΣΕΦΙΚ αλλά και με την γυρομέτο, που αφορά τα μέταλλα και τα μη σιδηρούχα μέταλλα, ε, τη σχετική βιομηχανία και με την Κονκάβε που είναι η Ευρωπαϊκή Πετρελαϊκή Βιομηχανία χερσαία βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου, ε, δεν, αυτό που κάνουμε μαζί τους ε, δεν είναι εργασίες ε, συμμόρφωσης. Πρώτον, υπάρχουν κάποια ζητήματα επιστημονικά δύσκολα, οι πετρελαϊκές ροές, είναι μείγματα χιλιάδων χημικών και τίθενται διάφοροι κίνδυνοι όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου και τη δοκιμή τους και η βιομηχανία αξιολογεί και τεστάρει αυτά τα χημικά Ω προ τον κινδυνό του εδώ και χρόνια και εμεί ε, συζητήσαμε μαζί του το πώ το βλέπουμε εμεί ε, ώστε βάσει τη δική τους εμπειρία να αποφασίσουμε εμεί, όχι μαζί με αυτού, εμεί να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τι άλλο κάνουμε σε τέτοιε συζητήσει. Μοιάζει με αυτό που κάνουμε όταν καθόμαστε κάτω με τούντε ε, για οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Πριν κάνουν την αίτησή του, εξηγούμε τη δική μα εμπειρία. Πότε μπορούν να κάνουν μία δήλωση εξαίρεση σε αποδοκιμές και ποτέ όχι για παράδειγμα. Είναι νωρίς λοιπόν ε, ε, αυτή η βοήθεια που παρέχουμε, αλλά τους βοηθάμε για να λάβουμε έναν καλύτερο φάκελο. Τους εφιστούμε την προσοχή στο τι μας βρίσκει να διαφωνούμε όσον αφορά τους φακέλους τους και τη συμμορφωσή τους, αντί να σπαταλάμε χρόνο σε επίσημες διαδικασίες να εξηγούμε πράγματα τα οποία τελικά καταλήγουν να ε, συμμορφώνονται. Κερδίζουμε δηλαδή σε αποτελεσματικότητα. Απλά αποτελεί ε, μια κατάσταση στην οποία ανταλλάσσουμε ε, πληροφορίες, γνώσει, εμπειρία, αλλά όχι παράλληλα πολύ πριν ξεκινήσουμε τη ρυθμιστική δράση. Ελπίζω όλα αυτά να εξήγησαν καλύτερα τις ανησυχίε μου. Είμαι έτοιμος ε, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας και δεν πρόκειται να αρχίσω να κρύβομαι αν κάτι ξέχασα να απαντήσω ευχαρίστως να το ξαναδούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη, λεπτομερέστατη και ειλικρινέστατη απάντηση και αντίδρασή σας στα σχόλια των συναδέλφων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ε, δεν ξέρω, αν θέλετε να ξαναπάρτε το λόγο τώρα, ε, μην μακρηγορήσετε, αν έχετε και άλλες ερωτήσεις και άλλες αντιδράσεις. Υπάρχει η ευκαιρία να συζητηθούν ε, αυτά τα θέματα και εκτός της σημαίνει συνεδρίαση, σε άλλο πλαίσιο, να συνεχίσετε τις επαφές. Αλλά θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Έικχουτ και στην κυρία Ριβαζή για να κάνουν κάποια σχόλια ή ερωτήσεις και μετά στον κύριο Χάνσεν για να τις απαντήσει. Κύριο κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομο θα είμαι. Σας ευχαριστώ κύριε Χάνσεν για την απάντησή σας και πιστεύω ότι αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να κάνουμε ακριβώ γιατί είναι πράγματι ανησυχητική. Θέλω όμως να δώσω μια συνέχεια ε, ε, ε, στα νούμερα. Είπατε ότι κάνατε ελέγχου συμμόρφωση για 700 φακέλους που δεν είναι 5% αλλά πηγαίνει προς την κατεύθυνση ε, του 5%. Αλλά τα δύο τρίτα των όσων ελέγξατε δεν συμμορφώνονται. Και συζητάμε για πολύ ανησυχητικέ ουσίες στο REACH, αλλά ε, προηγουμένως θα πρέπει να συμμορφώνεται ο φάκελος, αλλιώς δεν θα πρέπει να κυκλοφορεί το προϊόν στην αγορά. Αν τα δύο τρίτα των όσων ελέγξετε δεν είναι ως τα όφυλα, τι στόχο έχετε για το χρόνο, όταν θα ξανάρθετε εδώ, ε, έχετε κανένα στόχο για το πόσοι φάκελοι που δεν είναι ε, σε συμμόρφωση και όσοι παραμένουν μετά από ένα χρόνο, τι θα τους κάνετε, θα υπάρξει καμία κύρωση. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι υπήρξε μια επιλογή για το μοντέλο. Ε, δηλαδή πρώτα καταχώρηση όπως γίνεται με τα φάρμακα ε, και έγκριση και κυκλοφορία στην αγορά. Ε, μας είπατε ότι είχατε μεγάλη καθυστέρηση. Εντάξει, ε, το δέχομαι αυτό για τις χημικές ουσίες, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, κάθε βιομηχανία που εισάγει στην αγορά όχι χίλιους τόνους που ήταν ένα τόνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι και ε, εγκεκριμένη. Αλλιώς τι εγγυήσεις έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι δεν θα υφιστάμεθα τοξικές χημικές ουσίες. Με τη σημερινή διαδικασία δεν υπάρχει εχέγγυο προστασίας της δημόσιας υγείας. Και μας λέτε ότι δεν έχουμε χρόνο να τα ελέγξουμε κτλ. Και, και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Μα αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε εκτεθειμένοι στη ρήπανση των χημικών ουσιών και με την υγειονομική κρίση που ζούμε. Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε ότι από εδώ και μπρο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η έγκριση για να κυκλοφορήσει. Και για το θέμα της απαγόρευσης. Διαπιστώνεται, ας πούμε, ότι ένας φάκελος δεν συμμορφώνεται. Και τελικά δεν συμμορφώνονται με το ΡΙΤΣ. Οι εθνικέ αρχέ είναι εκείνε που είναι αρμόδιε για τα μέτρα εκτέλεση. Δηλαδή, βγαίνετε εσεί όπου είστε ο ΕΧΑ και λέτε ο φάκελο δεν είναι πλήρη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πούν να απαγορεύουμε την κυκλοφορία τη ουσία αυτή. Αυτό είναι. Μπορείτε λίγο να μα το διευκρινίσετε το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριο Πιέχα και πάλι ε, είχε ζητήσει το λόγο για να κάνει κάποιες ερωτήσεις και σχόλια πριν επανέλθουμε στον κύριο Χάνσεν για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να σας πω ότι <laughs> μου δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά. Ε, χαίρομαι που είστε εδώ και είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε στη συζήτηση με μεγάλη ε, ειλικρίνεια. Ε, πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε ο οργανισμός να έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Για μένα το σημαντικότερο ποιο είναι η αξιοπιστία. Έχουμε τους κανονισμούς αυτούς, το REACH και άλλους, αλλά θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι στα μάτια των πολιτών μας. Εγώ δεν εκπροσωπώ εμπειρογνώμονες, Ευρωπαίους πολίτες εκπροσωπώ που με έχουν ψηφίσει και ο κόσμος ανησυχεί. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα φυτοφάρμακα, για την αποθήκευση των αποβλήτων και όλα αυτά. Ο κόσμος ανησυχεί για αυτά τα θέματα. Ερώτηση, μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα περισσότερα ε, για κάτι που απασχολεί πολλές χώρες και δυστυχώς και την Πολωνία. Πώς αποθηκεύονται τα τοξικά προϊόντα και τα τοξικά απόβλητα. Τι γίνεται με τη διάθεση των τοξικών αποβλήτων. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορεί η Ευρώπη να εξάγει ε, δηλητήρια σε τρίτες χώρες, γιατί δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, το μετατοπίζει. Ευχαριστώ και πάλι και καλή τύχη στην αποστολή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Χάνσεν. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από την τελευταία παρέμβαση και σας Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, πράγματι, αξιοπιστία, ε, εμπιστοσύνη και η διαχείριση των αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σαφώς ηγετικό ρόλο ε, όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται σε διεθνέ επίπεδο. Βέβαια, το θέμα τελικά είναι τα νούμερα. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομούμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, αλλά και ένα διεθνές ε, θεματολόγιο για την διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αποβλήτων. Πράγματι αποτελεί τη βάση για τις εργασίες μας με δύο τρόπους μάλιστα. Εάν δεν είμαστε αξιόπιστοι, στα μάτια των ψηφοφόρων, τότε σίγουρα δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που την κάνουμε. Από την άλλη, αν το καταφέρουμε αυτό, τότε πράγματι προστατεύουμε τους πολίτες. Είναι κριτικό το μάτι του ε, ψηφοφόρου και αν μπορούμε να ικανοποιήσουμε ε, τον ψηφοφόρο, τότε κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ίσως θα πρέπει να προσθέσω ότι όπως βλέπω εγώ τις εργασίες ε, του ΕΧΑ και ε, η μικρή σφραγίδα που θέλω να βάλω εγώ στη μεγάλη σελίδα ε, είναι... Για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη και την αξιοπιστία τη δική μας, θέλουμε οι οι πολίτε να δουν ότι γινόμαστε όλο και πιο αποτελεσματικοί στι εργασίες μας, ε, δηλαδή ότι δαπανούμε καλά τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το άλλο θέμα είναι η συνέπεια που ήταν και ένα από τα θέματα στην συζήτηση για τη γλυφοσάτη. Εκεί αναφέρθηκε η ασυνέπεια και η αβεβαιότητα. Μπορώ όμως να σας... Ε, θα μπορούσα και να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα αν είχαμε το χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε άλλες περιπτώσεις όπου υπήρξαν ασυνέπειες. Για πολύ καλούς λόγους ε, που όμως είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε την αξιοπιστία και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη είναι το θέμα των συνεργειών. Ο ΕΧΑ έχει την δυνατότητα έχει τις απαραίτητες δεξιότητες ε, για να επιδιώξει τις συνέργειες αυτές ε, και να αναλάβει ε, περαιτέρω καθήκοντα στο πλαίσιο των χημικών. Όσον αφορά τα απόβλητα, ασχολούμαι τα χημικά εδώ και 30 χρόνια. Όπως σας είπα, ε, τα χημικά είναι το πάθος μου. Ε, βλέπω τον κόσμο ε, μέσα από τα χημικά. Βλέπω σε αυτή την αίθουσα τα χημικά που υπάρχουν, πέρα από κάποιες οργανικές ουσίες. Αλλά, εν πάση η πολιτική χημικών και η πολιτική αποβλήτων για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Απλά στο θέμα των αποβλήτων ο κόσμος ε, εξετάζει κάθε πράγμα σαν ένα αντικείμενο, ενώ εγώ το βλέπω σαν συνδυασμό χημικών. Για μένα λοιπόν αυτές οι δύο πολιτικές είναι ε, ένα πράγμα και γι' αυτό η ε, πολιτική για την κυκλική οικονομία είναι πολιτική για τα χημικά. Όσον αφορά την αποθήκευση δηλητηρίων, τοξικών ουσιών, αν ε, εννοείται την ε, αποθήκευση ε, αποβλήτων, τότε αυτό σίγουρα είναι θέμα αποβλήτων, αλλά οι γνώσεις και οι τεχνολογίες σίγουρα είναι θέμα του τομέα των χημικών. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις ουσίες αυτές. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί εδώ η, η γνώση μας και οι δεξιότητές μας. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα νούμερα, ναι, φυσικά θέλουμε να ε, αυξηθούμε. Σε 12 μήνες ε, μπορεί να ε, με παραπέμψετε στα λόγια που λέω σήμερα. 10 χρόνια, 10 μήνες βρίσκομαι στη θέση αυτή και θα φτάσει η ώρα που θα μπορούμε να πούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Πάντως αυτό που προσπαθώ εγώ και το προσωπικό επίσης του ΕΧΑ είναι ότι θέλουμε να βρούμε τα πιο σημαντικά χημικά όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και συχνά ε, η δουλειά πάνω σε μία χημική ουσία είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι για κάποια άλλη. Δεν θέλω να αποθαρρυνθεί το προσωπικό του ΕΧΑ όσον αφορά την ανάληψη μιας δύσκολης υπόθεσης και να αναλάβει κάποια άλλη πιο εύκολη για να έχουμε καλύτερες στατιστικές. Από την άλλη, σίγουρα θέλω να κάνω πολλή δουλειά και προσπαθώ να συνδυάσω αυτά τα δύο. Δεν ε, το έχω καταφέρει ακόμα με το προσωπικό που έχω στη διάθεσή μου. Σε 12 μήνες όμως, ρωτήστε με πάλι σε ποιου τομεί έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. Δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή ε, να κάνω περισσότερα. Θα κάνουμε περισσότερα, θα καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στο θέμα της συμμόρφωσης. Το πώς θα φανεί αυτό ε, στις στατιστικές, ως αριθμός θεμάτων δηλαδή, ε, αυτό θα φανεί. Αυτή τη στιγμή 200 υποθέσεις το χρόνο εξετάζουμε και μάλλον προχωράμε σε 200 ουσίες το χρόνο. Βλέπουμε δηλαδή επιτάχυνση και ε, εντατικοποίηση των προσπαθειών μας. Εάν όμως βρούμε 200 ουσίες που να καλύπτουν το 30% τα 100 του όγκου στην αγορά, τότε θα είναι καλύτερο από το να κάνουμε 300 ε, ουσίες οι οποίες να καλύπτουν πολύ μικρότερο ποσοστό της αγοράς. Ε, του χρόνου θα σας πω πώς μπορούμε να μετρήσουμε τις επιτυχίες μας ε, και θα μπορέσω να σας δείξω ε, σε ποιους τομείς έχουμε βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και για τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο που είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Όσον αφορά τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, ε, θα συνεδριάσουμε στις 12 Νοεμβρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, και κατόπιν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, σε δύο εβδομάδες από τώρα. Έτσι φτάνουμε στο τέλος ε, της ε, σημερινής μας ε, συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας ευχαριστώ που συμμετείχατε ενεργά στη συζήτηση. Λήξη της συνεδρίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Sorry. Yeah, but, um, well,